Ο Πρόεδρος. Καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε. Σας χρωστώ μια εξήγηση, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Χέρινς ε, Γκαρθία θα έρθει πολύ σύντομα. Η πτήση της καθυστέρησε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν είναι ακόμα εδώ. Ο κύριος Αχμή πάλι είναι σε μια άλλη συνεδρίαση. Οπότε θα περιμένουμε νομίζω μέχρι τις 3 και στις 3 θα αρχίσουμε την συνεδρίασή μας και θα ζητήσουμε από την κυρία Μίρα να πάρει το λόγο. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να καλωσορίσω εδώ τους νέους προσκεκλημένους μας. Είναι νέοι Γεωργοί από την Ολλανδία που έχει καλήσει και η κυρία Σφάγερ και βλέπετε το μπλουζάκι μου έτσι. Μόνο που μικραίνουν τα τίσερ το τελευταίο καιρό, δεν ξέρω, και με στενεύει. Τι να κάνουμε. Κύριε Σράιερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια ομάδα νεαρών ε, αγροτών από την Ολλανδία μαζί μας από τις σχετικές οργανώσεις ε, και ενώσεις νεαρών αγροτών και είναι πολύ σημαντική λοιπόν η μέρα. Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσο μπορούμε να παραμείνουμε αγρότες στην Ευρώπη και σίγουρα ε, μετά τη νέα αγροτική και πολιτική. Κάθε χώρα είναι διαφορετική και κάθε χώρα έχει διαφορετική δυναμική. Αλλά σήμερα λοιπόν είναι στα πίσω έδρανα και μιλώ όχι εξ ονόματα δικό μου, αλλά και του κυρίου Χάιτομα που κάθεται πίσω Σε όλη αυτή την λοιπόν θέλουν να ξέρουν και θέλουν να του πει η Ευρώπη πού οδεύουμε. Γιατί συχνά λέμε ότι δεν υπάρχουν νέοι αγρότε. Μα κοιτάξτε, έχουμε αρκετού νεαρού αγρότε εδώ μαζί μα στην αίθουσα. Αλλά γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η νέα γεωργική πολιτική. Θα πρέπει να είναι βιώσιμη, αποτελεσματική και εφικτή, με πιο ε, λίγου κανόνε, αλλά να μπορεί και ο αγρότη να παραμείνει αγρότη. Σα εύχομαι λοιπόν μια καλή συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας αυτή. Ας δούμε λιγάκι τα άλλα τα συνηθισμένα ε, σημεία στην ημερήσια διάταξη αναμένοντας τους συναδέρφους. Δεν ξέρω αν πιστεύετε στην κλιματική αλλαγή αλλά νομίζω ότι εδώ από πρώτο χέρι μπορείτε να διαπιστώσετε τις κλιματικές αλλαγές που έχουμε από ώρα σε ώρα εδώ στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε πρώτα απ' όλα. Ωραία. Σημείο 2. Μεταδίδεται στο διαδίκτυο η σημερινή συνεδρίασή μας και έχουμε μαζί μας και έναν δημοσιογράφο από την Αυστραλία. Γιατί βλέπετε κάθε χρόνο η η αντιπροσωπεία των ε, χορηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αυστραλία μαζί με την Qantas απονέμουν κάθε χρόνο ένα βραβείο σε Αυστραλό δημοσιογράφο. Είναι το βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Qantas για να μπορεί ένας δημοσιογράφος να έρθει στις Βρυξέλλες και σε κάποια άλλη χώρα μέλος. Έτσι εξοικειώνονται με τα ευρωπαϊκά ζητήματα και μπορούν ε, τα ευρωπαϊκά ζητήματα να τα μεταφέρουν στους συμπατριώτες τους στην Αυστραλία αργότερα. Φέτος λοιπόν έχουμε μαζί μας ε, τον κύριο Μπρέτ Worthington, ο οποίος ασχολείται με τα θέματα της υπαίθρου και της γεωργίας. Δουλεύει για το ABC που είναι ε, το Αυστραλιανό δίκτυο τηλεόρασης και ένα από τα κύρια μέσα ενημέρωση Αυστραλίας. Είναι μαζί μας λοιπόν. Σήμερα θα μαγνητοσκοπήσει αυτή τη συνεδρίαση. Μην αναφέρετε ότι αργήσαμε να αρχίσουμε, λέει ο πρόεδρος στον κύριο Βέρθιγκτον. Αλλά βέβαια εντάξει, ξέρω ότι αφού το λέω, σίγουρα θα αναφερθεί. Τι να κάνουμε. Καλώς ήρθατε πάντως. Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε ε, μαζί, μαζί μας σήμερα. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες και δεν έχουμε στα τσέχικα, ε, μαλτέζικα, σλοβάκικα και γκέλικ. Μήπως να αλλάξουμε τη σειρά των θεμάτων στη συνεδρίαση, αν και βέβαια είναι ένα πακέτο και θα ήταν καλό να αρχίζαμε με την παρουσίαση της κυρίας Χέρανς Γκαρθία θα ήταν η λογική σειρά να εξετάσουμε τις εκθέσεις που έχουμε να εξετάσουμε σήμερα. Αλλά τι να γίνει, θα αρχίσουμε κάπως διαφορετικά. Θα αρχίσουμε από το επόμενο θέμα που είναι η διαχείριση, ο έλεγχος της ΚΑΠ. Η συγκεκριά μας είναι η κυρία Μίλλερ και έχουμε γνωμοδοτήσεις από την DEVE, INTA, Budget Κοντ και όπως γίνεται και με τους οριζόντιους κανονισμούς κάθε φορά, έχουμε διαπραγματεύσεις, έχουμε 863 τροπολογίες και η συνάδελφος, η κυρία Μίλλερ, σίγουρα θα μας πει περισσότερα. Έχουμε όμως γνωμοδότηση τελικά μόνο από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Αναμένουμε όμως και η Ρέγγι και η Κοντ και η Ντέβε θα υιοθετήσουν τις δικές τους γνωμοδοτήσεις πριν από τις 7 Φεβρουαρίου. Φέτος, ε? το τονίζω και αυτό, λέει ο Πρόεδρος. Γιατί πραγματικά Του παίρνει πολύ χρόνο να ετοιμάσουν τι γνωμοδοτήσει τους. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ πέρα όλους μας τους προσκεκλημένου. Σε αυτό το σημείο λοιπόν τη ημερήσια διάταξης, στο σημείο 4, ξέρω ότι ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής θα είναι μαζί μας. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε και να αρχίσουμε ζητώντας και πάλι συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αν είναι έτοιμη κυρία Μίλλερ, παρακαλώ. Είναι έτοιμη η συγκήτρια. Οπότε παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Μίλλερ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, θα ήθελα κι εγώ να ξεκινούσαμε πρώτα με τα στρατηγικά σχέδια, αλλά στην περίπτωση αυτή να σας ανακοινώσω ποιες είναι οι προθέσεις μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις διαφανείς συνθήκες, σε ό,τι αφορά την δίκηση. Αυτές ήταν οι προτάσεις μου λοιπόν στην έκθεση του Νοεμβρίου σε ό,τι αφορά τον ε, οριζόντιο κανονισμό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία η οποία έχει πραγματικά με έχει χαροποιήσει με τους σκιώδεις και μπορώ λοιπόν να σας ενημερώσω για το τι έχει συμβεί. Έχουμε, είχαμε 163 τροπολογίες, είχαμε 4 τεχνικές συνεδριάσεις ως τώρα. 863, συγγνώμη, τροπολογίε και μάλιστα μια τελευταία τεχνική συνάντηση σήμερα το πρωί. Από οριζοντίας απόψη, αυτός ο κανονισμός λοιπόν έχει σημεία επαφή και με τι τρει νομοθετικέ προτάσει σε ό,τι αφορά τα νέα στρατηγικά σχέδια που αναπτύσσονται, τι άμεσε πληρωμέ και την ανάπτυξη τη υπέτρου. Το άρθρο 121 των στρατηγικών σχεδίων είναι αυτό το οποίο αναφέρεται πιο συχνά στην, στον οριζόντιο κανονισμό. Η βασική αρχή για την επιτευξη των συμβιβασμών είναι να εστιαστούμε πρώτα στα σημεία κλειδιά και καταρχάς να αποφασίσουμε το σύνολο με τους σκιώδεις συζητητές και μετά να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια κοινή κατεύθυνση και στη συνέχεια να υποβάλουμε προτάσεις για το τι είναι εφικτό ή όχι. Εξετάζοντας ε, άνθρωπος προς άθρο το θέμα αυτό, όπω κάνουν οι συνάδελφοι, δεν θεωρώ ότι έχει νόημα εδώ στον οριζόντιο κανονισμό, γιατί πολλά είναι αλληλεξαρτώμενα. Υπάρχουν επίση πάρα πολλέ ε, συνδέσει με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώ και με τον κοινό κανονισμό, το κανονισμό για τι κοινέ διατάξει. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξουμε συνολικά. Έχουμε συζητήσει τα εξή σημεία ω τώρα. Ένα σημείο αρχή, το οποίο συζητήσαμε και σήμερα πολύ εντατικά. Είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην γενική της μορφή. Ξέρετε ότι βασίζεται στην τήρηση των κανόνων το θέμα της συμμόρφωσης. Το μελλοντικό σύστημα λοιπόν θα πρέπει να βασίζεται πιο πολύ σε επιδόσεις, σε performance. Μία λοιπόν ξαφνική αλλαγή από το σημερινό σύστημα στο σύστημα απόδοσης θεωρώ ότι δεν θα λειτουργήσει. Είμαστε απόλυτα πεπισμένοι γι' αυτό. Και το συζητήσαμε αυτό και σήμερα πάλι και πιστεύω προσωπικά ότι αποτελεί αυτό ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση το οποίο προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό όμω που πρέπει να διατηρηθούμε είναι πώς μπορούμε να διαρθρώσουμε καλύτερα το σύστημα αυτό, πώς μπορούμε να πληρώσουμε και τις προδιαγραφέ ε, περί απόδοση και να διατηρήσουμε τη βάση τη γνωστή για τους αγρότες. Αναγκαστικά θα υπάρξουν ε, παράλληλα συστήματα προκειμένου να υπάρξει μετάβαση σε ένα σύστημα που θα βασίζεται στην απόδοση. Η δική μου η εκτίμηση που βασίζεται και στην πρακτική μου εμπειρία είναι η εξή. Έχουμε το παλιό σύστημα και έχουμε και στο... στη μελλοντική πολιτική αυτή και μια μεταβατική ε, ρύθμιση η οποία θα μας οδηγήσει τελικά σε ένα σύστημα απόδοσης στην επόμενη φάση την οποία και επιθυμούμε να πετύχουμε. Σκοπός μου είναι να ψηφιστεί τελικά ένα κείμενα για την ε, γεωργία που ε, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια των σχετικών διοικητικών υπηρεσιών και ε, τη μέγιστη ευελιξία για τις λήψεις αποφάσεων. Φυσικά μπορούμε να πούμε ότι όλοι αυτοί οι δείκτες που καθορίζονται στο μέλλον θα είναι πιο λίγοι από αυτούς που έχουμε σήμερα. Αλλά μιλάμε για μεγάλη διαφορά κατά πόσον ε, θα παραμείνουμε στο τρέχον σύστημα με τις σχετικές διατάξεις ε, που πρέπει να πληρώνονται όλες τους με 250 ε, προδιαγραφές ή κατά πόσον θα βασιζόμαστε στο μελλοντικό σύστημα όπου θα υπάρχουν πραγματικά μετρήσιμα αποτελέσματα σε σχέση με την απόδοση. Αυτό θεωρώ ότι θα κληθούμε να το συζητήσουμε και να το αποφασίσουμε και θα πρέπει να στήσουμε λύσεις με τους κοιόδες εισηγητές. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το θέμα της, ε, του αποθεματικού για την κρίση. Είχαμε πάνω από 50 τροπολογίες για το θέμα αυτό. Με διάφορε αξιώσει ό,τι αφορά τα χρήματα που θέλουν, για παράδειγμα, μερικοί να μείνουν εκτό του ΠΔΠ ή εντό του ΠΔΠ. Άλλοι κάποιοι θέλουν να μείνουν εκτό ε, τη ε, του προπολογισμού για την κοινή αγροτική πολιτική. Άλλοι θέλουν να μείνουν εντό. Θέλουμε να υπάρχει μια ξεχωριστή, ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο, ένα ξεχωριστό φάκελο ω αποθεματικό κρίση και να υπάρχει και δυνατότητα παρέμβασης σε κανονικές ε, διακυμάνσεις της αγοράς. Αυτές λοιπόν είναι πολλές και διαφορετικές απόψεις και σε καιρούς όπου είναι όλο και πιο πιθανές οι κρίσεις, είναι σημαντικό να έχουμε μια σωστή ΚΑΠ με σωστή πρικοδότηση και εύρυθμα λειτουργούσα πολιτική που να μπορεί πραγματικά να παρέμβει σε περίπτωση ανάγκης και κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω να υπάρχει αποθεματικό κρίσης, αποκλειστικά όμως για κρίσεις, όχι για παρεμβάσεις στην αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καταρχάς τους συναδέλφους για τα σχόλια που κάναν, για την καλή συνεργασία. Άψογη υποστήριξη στα πλαίσια από την ε, γραμματεία μάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε διευκρινίσει και τη πολλά ζητήματα και έχουμε κάνει μεγάλα βήματα σε ό,τι αφορά την επιτευξή συμβιβασμών. Το θέμα λοιπόν είναι πραγματικά να υπάρχει διαφάνεια σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, η μέγιστη απλοποίηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει από τους φιλελεύθερους ε, ένα σεμινάριο σε ό,τι αφορά και αυτούς τους δείκτες, προκειμένου να έχουμε ενδεχομένω ε, πιο σαφείς απόψεις από πλευράς και των εμπειρογνωμών. και νομίζω ότι όλοι θα προσκληθούν στην εκδήλωση αυτή. Θα προσκληθεί μάλλον το σύνολο της Επιτροπής και είμαι βέβαια ότι τελικά θα καταφέρουμε να επεξεργαστούμε και να καταλήξουμε σε μία ισχυρή τοποθέτηση. Παρ' όλα αυτά λοιπόν γίνονται προτάσεις οι οποίες επεμβαίνουν στη στρατηγική, στα σχέδια στρατηγικής και εδώ θα πρέπει να κάτσω να συζητήσω κατά πόσον ε, μπορούμε ξανά να ανοίξουμε θέματα περί στρατηγικής στον οριζόντιο κανονισμό, γιατί τα υπόλοιπα θέματα είναι όλα επιτάπητος. Και νομίζω ότι πραγματικά θα καταφέρουμε να εργαστούμε και τάχιστα. Να βρούμε καλές ε, θέσεις και τελικά να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και στο μέλλον με πιο ισχυρή τοποθέτηση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Αν θα μπορούσατε να μας δώσετε και την ημερομηνία των σεμιναρίων αυτών, ώστε να τα σημειώσουμε. Και μετά, σκιώδες συζήτητες, δεν θέλω να σας περιορίσω, μεν, αλλά σας παρακαλώ σε τρία λεπτά να κάνετε τις παρεμβάσεις. Τέλος πάντων, με κάποια ελαστικότητα. Ο κύριος Νταντάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για το έργο της. Δουλέψαμε πολύ μαζί. Και είναι αλήθεια ότι κάποια σημεία δεν δημιουργούν προβλήματα και τα δύο σημεία στα οποία αναφέρθηκε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και δημιουργούν αποκλίσεις μεταξύ των ομάδων. Θα αρχίσω από το δεύτερο, που ίσως είναι και το πιο εύκολο, αυτό το αποθεματικού. Εξάλλου τίθεται και το θέμα του όρου. Αποθεματικό είναι ο σωστός όρος, ώστε να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και σύγχυση. Αυτά τα, τα χρήματα λοιπόν που διαχωρίζονται χρησιμεύουν σε περίπτωση μεγάλων κρίσεων όπως εκείνη του γάλακτος του 2016, την κλιματική ή είναι μια γραμμή στον προπολογισμό η οποία χρησιμεύει ώστε κάθε χρόνο με τα διάφορα συστήματα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιούνται. Το διαχειρίζεται όλο και λιγότερο, αλλά πάντως το διαχειρίζεται ακόμα. Αυτό το κονδύλιο πρέπει να είναι ενιαίο ή μπορεί να χωρίζεται. Πρέπει να είναι στις γεωργικές πιστώσεις ή εκτός αυτών. Κρίσεις δεν έχουμε μόνο στη γεωργία και ο κίνδυνος είναι αν έχουμε μια γραμμή κρίση που να εγγράφεται κάπου αλλά να μην είναι πραγματικά στον προπολογισμό της Γεωργίας, τότε με οποιαδήποτε κρίση προκύψει στην Ευρώπη θα τα χρησιμοποιήσουμε. Το γεγονός λοιπόν αν δεν έχουμε χωριστή γραμμή με τον καιρό, κινδυνεύουμε να μην έχουμε αρκετά χρήματα στο αποθεματικό για τις μεγάλες κρίσεις. Βλέπουμε την αδυναμία αντίδραση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που οφείλεται στην αδυναμία του προπολογισμού. Ξηρασία φέτο, για παράδειγμα. Ε, δεν έκανε τίποτα τελικά η Ευρώπη κοινοτικά, ενώ η Γεωργία είναι ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα λίγα διαθέσιμα κονδύλια που υπήρχαν, αν τα είχαμε ε, μοιραστεί, είχαν μοιραστεί ανάμεσα στους δικαιούχους που υπέφεραν από την ξηρασία, ψίχουλα θα παίρνανε. Θα ήταν ντροπή. Το αποθεματικό αυτό λοιπόν πρέπει να είναι καλά περικοδοτημένο και να επιστρέφονται τα χρήματα τα οποία δεν έχουν δαπανηθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Τώρα το άλλο που ανέφερε και η κυρία Μίλλερ, που έχει να κάνει με τα διαφορετικά συστήματα ελέγχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει να εγκαταλείψουμε το σύστημα της ε, τεκμηρίωσης της εποπτείας που καθορίζεται από τα κείμενα και η κάθε χώρα να κάνει όπως θέλει και να ελέγχει ό,τι εκείνη θέλει. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε διαφορετικούς δικαιούχους από χώρα σε χώρα. Άρα αρχίζει μια επανεθνικοποίηση με αυτόν τον τρόπο. Και έπειτα αυτό το οποίο μας προτείνεται είναι να έχουμε έλεγχο επιδόσεων. Ο όρος επιδόσεις δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλο, γιατί αυτό που προτείνει ουσιαστικά είναι να ελέγχουμε ότι αν είπαμε ότι θα έχουμε 100.000 εκτάρια βιολογική καλλιέργεια, πρέπει να είναι 100.000 εκτάρια. Και αν δεν είναι, πρέπει να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε γιατί δεν είναι. Ε, δεν πάει και πολύ μακριά αυτό. Σε κάποιε ομάδε θέλουν να πάνε πολύ μακριά και να κάνουν την ε, πολιτική γεωργίας κάτι άλλο από την πολιτική γεωργίας, να την κάνουν περιβαλλοντική πολιτική. Συμφωνώ για τη διάσταση του περιβάλλοντος μεν, αλλά διαφωνώ στο να αφαιρεθεί ο χαρακτήρας ε, της γεωργίας από αυτή τη συζήτηση. Είναι περίπλοκο το θέμα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάποιες διευκρινήσεις κάθε τόσο. Οι όροι δεν είναι σαφείς οδηγούν σε σύγχυση. Στο λίγο χρόνο που μας μένει, μέχρι το Μάρτιο που πρέπει να ψηφίσουμε εδώ, καλό θα ήταν αυτά να αποσαφιστούν. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρος. Ο κύριος Σεροσάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω για όλα αυτά τα τόσο άρτια που μας είπε η κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ και για τη συνεργασία. Ε, είμαι ο σκιώδης εισηγητής. Ε, υπήρχαμε κάποιες ε, διαφωνίες, αλλά τελικά συνεργαστήκαμε επικοδομητικά, γιατί υπήρχε θετικό πνεύμα. Είναι πάρα πολύ τεχνικό αυτή η έκθεση. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις κυβερνήσεις και στην εξέλιξη της ΚΑΠ βλέπουμε ότι το θέμα είναι η επιδόση τα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση που χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε, να τη συζητήσουμε περισσότερο, να δούμε πώ θα βρούμε όσο γίνεται καλύτερε λύσει για όλο τον κόσμο και του πολίτε και του γεωργού. Βλέπουμε τώρα, π.χ. διακρίνουμε κάποιου ε, κινδύνους, περισσότερη γραφειοκρατία, να βαρύνουν περισσότερο οι εθνικές ε, δημόσιες υπηρεσίες. Και υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και για τους γεωργούς, άρα θα πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει με τις τροπολογίες που αφορούν αυτά τα σημεία. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα κριτήρια, τους δείκτες, θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή στις διαφορετικές παρεμβάσεις, την πραγματικότητα στη, της γεωργίας. Έτσι να δούμε πώς θα υπάρχει ένας ε, κανονικός που είναι, ε, κανονισμός που είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Κάτι άλλο το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη είναι να βρούμε μια κοινή βάση. Αυτή να είναι τόσο στεγανή, ε, εκεί να βασίζονται όλα να είναι δίκαιη η ρύθμιση όσον αφορά την υλοποίηση της ΚΑΠ. Και αυτό να αφορά όλες τις εκμεταλλεύσεις. Και έτσι να μπορούμε να καλύψουμε την πολυμορφία που υπάρχει και επομένως να μην έχουμε επανεθνικοποίηση. Όσον αφορά τώρα το αποθεματικό της κρίσης, ε, το ανέφεραν άλλοι, ε, έχουμε το πρόγραμμα πλαίσιο, έχουμε μια προσωρινή ρύθμιση και κάλυψη από τον προϋπολογισμό και έχουμε πει ότι θα πρέπει ε, να υπάρξει κάλυψη από επιπλέον ποσά από έναν έκτακτο προϋπολογισμό για την περίοδο 14-20 είχαμε πει τώρα η αρχή του rollover θα πρέπει να προσαρμοστεί επίσης σε αυτές τις ρυθμίσεις. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κατάινεν, έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ. είναι σε καλά χέρια το θέμα και ευχαριστώ την εισηγήτρια γιατί αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση θα καλυφθεί από τρεις κανονισμούς. Σας ε, τονίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε, θα πρέπει να συντονίσουμε τις ευμέρους προτάσεις και έτσι το Κοινοβούλιο να έχει τις διαβροντές που θα έρθουν συνεπή κρυστάλλινη θέση και Ελπίζουμε έτσι να δουν το θέμα και οι εισηγητές. Να λιάνουμε τις διαφορές, να έχουμε κάποιες προτεραιότητες, να βοηθήσουμε τους παραγωγούς και να απαλλαγούμε από την γραφειοκρατία. Τώρα όσον αφορά την ερεσιμότητα, να λάβουμε υπόψη την επικουρικότητα Να δούμε τι θα γίνει με το νέο μοντέλο. Να μην υπάρχει πανεθνικοποίηση, μην υπαγορεύεται ότι θα γίνει το κράτος μέλος. Και να μην έχουμε επίσης επικάλυψη των, των εργοδιών των αριθμιστικών αρχών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή άτυπα αναγνωρίζει ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα είναι λογικό βήμα, αλλά αυτή η πρόταση ουσιαστικά επιμένει στην σύστημα που υπάρχει, να μην δίνονται λεφτά και να μην ε, αναλαμβάνονται ρίσκα. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως. Ε, τι θα κάνουμε, θα πούμε δηλαδή στα κράτη-μέλη ε, που δεν τα πάνε καλά με τους κανόνες, θα τους δώσουμε ελεύθερο πεδίο. Δεν το θέλουμε αυτό. Κατά δεύτερον, θέλουμε να υπάρχει μια σιγουριά. Μια σιγουριά κυρίως ότι ό,τι αφορά τα διοικητικά, το διοικητικό αχθός γιατί οι τρέχοντες κανόνες ε, έχουν ε, λένε ότι θα πρέπει να επιστραφεί για τα τρίτη ταρτά οι επιδοτήσεις οι οποίες δεν τηρούν τους κανόνες. Στην πρόταση αυτή ε, το ποσοστό αυτό πάει στο 80%. Δεν μπορούμε να επιτηρήσουμε τα μέσα αυτά για τα κράτη-μέλη αν αφιερώνονται στο κλίμα και στο περιβάλλον. Γιατί αυτό λέει ο πρώτο πυλώνας. Είναι καλό να υπάρχουν οι πρώτε αυτέ, στον πρώτο πυλώνα, αυτά τα αυτή η πόρη και, και ο δεύτερος πυλώνας να παραμένει σε ό,τι αφορά τέτοιες συμφωνίες. Στο 3.1 υπέβαλα μία τροπολογία σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους, όπως είναι οι οργανώσεις οι οποίες έπραξαν καλή την πίστη. Για από αυτές λοιπόν να μην χρειάζονται να ζητάμε επιστροφή των ε, πόρων, γιατί έτσι δημιουργείται η δυσπιστία στους κανόνες και αποτρέπεται και η συμμετοχή και στα απορροκυπευτικά ισχύει αυτό, αλλά και άλλο. Και ελπίζω να μην υπάρξουν υπερβολικοί κανόνες, γιατί αυτό θεωρώ ότι θα αποτρέψει μια σωστή πολιτική, γεωργική πολιτική. Και ευχαριστώ και την κυρία Μούλερ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρε, Νομίζω ότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ κακή. Δεν συμφωνώ με την έκθεση ετήσιας επίδοσης που κάνει η πρόταση της Επιτροπής και γι' αυτό στηρίζω τον κύριο Νταντάν και τη δικιά του έκθεση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τρία χρόνια εκθέσεις επιδόσεων και αξιολογήσεις οι συμβαστικέ ε, τροπολογίες τώρα, δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω για αυτές. Πρώτον, οι προθεσμίες για τις εκθέσεις επιδόσεων. Είναι αδύνατον 15 Φεβρουαρίου να τα καταφέρουμε. Είναι αδύνατον για τις αρχές των χωρών μελών. Εγώ προτείνω την 30η Ιουνίου, αλλά έχω δει και άλλες προτάσεις που λένε 1η Ιουνίου. Εντάξει, θα μπορούσα να το δεχτώ και αυτό. Έπειτα, άρθρα 51 και 52 για την εκαθάριση λογαριασμών ετησίως. Αν υπάρχει ανταλλαγή μεταξύ χωρών μελών, οι προθεσμίες εδώ δεν θα έπρεπε να τροποποιούνται από κατεξουσιοδότηση πράξης. Μόνο από τους συνομοθέτες θα μπορούσαν να τροποποιηθούν, γιατί είναι πολύ σημαντικοί οι κανόνες αυτοί. Και αν οι οι πράξεις χρησιμοποιηθούν, τότε ούτε το Συμβούλιο, Ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να απορρίψει απαράδεκτα μέτρα. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριο Φλάνεγκαν. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σε σχέση με τις επιδόσεις, τις μετρήσεις επιδόσεων, φαίνεται να είναι μια εξαίρετη ιδέα, όμως στην πράξη δεν ξέρω αν θα είναι. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, έχουμε δει καταστάσεις όπου οι αγρότες κάνανε ό,τι έπρεπε να κάνουν, αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν και τόσο καλό. Σε εμά, στην περιφέρειά μου, για παράδειγμα, είχαμε ένα σε σχέδιο και μόνο 25% των στόχων επιτεύχθηκαν. Παρόλο που όλοι ε, ασχολήθηκαν και προσπάθησαν. Και οι υπηρεσίες ναι λένε ότι οι αγρότες έκαναν ό,τι μπορούσαν, από την άλλη μεριά όμως οι αγρότες παρά τη συνεργασία την καλή που είχαν δεν τα κατάφεραν. Τους ενδιαφέρει και η βιοπικιλότητα, έκαναν ό,τι τους ζητήθηκε. Τα αποτελέσματα όμως που πέτυχαν ήταν 25% αυτών που αρχικά αναμένονταν. Μα πρόκειται για πειράματα και οι αγρότες δέχτηκαν να συμμετάσχουν στο πείραμα. Το ότι δέχτηκαν να συμμετάσχουν στο πείραμα δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουν και 25% των αποδοχών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και ο κόσμος στρέφεται κατά αυτής της ιδέας. Οπότε, Πάρα πολύ ωραία ιδέα θεωρητικά, στην πράξη όμως είναι αλλιώ τα πράγματα. Ευχαριστούμε. Καλομπιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, το έχω πει και ξαναπεί. Η μεταρρύθμιση αυτή της κοινή ζωική πολιτική δεν είναι καλή. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε να γίνει χωρί καμία βεβαιότητα, χωρίς καμία βεβαιότητα σήμερα, δεδομένου του προπολογισμού τη ΕΚΑΠ για το 2020. Κανένας δεν λέει ότι μόνο κάποια ε, κονδύλια θα πάνε στους αγρότες. Τα άλλα θα πάνε είτε στην πολιτική διαχείριση των μεταναστών. Θα πρόκειται για ε, μετατόπιση των μεταναστών αυτών, όπου θα τους εγκαταστήσουμε στην Ήπεθρο ε, που ήδη υποφέρει. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε ιδέα τι ποσά θα φτάσουν στα χέρια των αγροτών μας ενώ θέλουμε να αποφασίσουμε με ποιο τρόπο θα τους τιμωρήσουμε αν κάνουν κάποια ασφάλματα στη χρήση αυτών των ακόμα άγνωστων ποσών. Οπότε, εύχομαι ότι καλύτερο σε όποιον θέλει να δοκιμάσει τέτοια πειράματα στους αγρότες μας και στις καλλιέργειές μας. Μα ακριβώ αυτοί οι αγρότες είναι που βλέπουν καθημερινά πόσο σκληρή είναι η Ευρώπη απέναντι στους ε, πιο αδύναμους, αλλά και πόσο χαλαρά αντιμετωπίζει τους πιο πλούσιους. Είτε πρόκειται για τη Βραζιλία, είτε πρόκειται για την Πολωνία, τα σφαγεία, οτιδήποτε. Η προτεραιότητα είχαμε πει ότι είναι η απλοποίηση. Προτεραιότητά μας όμως για όλους μας πρέπει να είναι να σώσουμε τη γεωργία των χωρών μας, γιατί από αυτό εξαρτάται η ανεξαρτησία στην διατροφή μας. Οπότε δεν βλέπω πώς μπορεί κανείς να υποστηρίξει επιτόπου αυτήν την ε, αλλαγή στην κοινή γεωργική πολιτική. Νομίζω ότι δεν πρέπει να τη λέμε κοινή γεωργική πολιτική, αλλά κοινή γεωργική τιμωρία. Ευχαριστώ. Κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σημαντικό το να συνειδητοποιήσουμε ότι για την ΚΑΠ Αυτά τα θέματα του, του δημοσιονομικά είναι πολύ σημαντικά και η σχετική πρόταση της Κομισιόν είναι σκανδαλώτης γι' αυτό το 15% ως περικοπή μέσα στα πλαίσια της γενικότερης αύξησης του κοινωνικού προϋπολογισμού. και με δεδομένο το Brexit και την αναθεώρηση που θα πρέπει να περάσουν τα μέτρα. Επομένω, θα πρέπει η Κομισιόν να διαβάσει στο κολέγιο των Επιτρόπων ότι αυτά τα μέτρα δεν θα περάσουν. Ε, γιατί έχει τόσα να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και η Γεωργία. Οπότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οτιδήποτε πόροι χρειάζονται για το αποθεματικό θα πρέπει να έρθουν από τον προϋπολογισμό που δεν αφορά την ΚΑΠ η γεωργία είναι μοναδικός τομέας που έχει προϋπολογισμό που τώρα θεωρείται ότι πρέπει να καλύψει και έκτακτα συμβάντα. Έχουμε σχετικές τροπολογίες. Αποθετικό, το, το αποθεματικό να προέλθει από αλλού, εκτός γεωργικού προϋπολογισμού. Τα είπαμε. Και σωστά είπαμε ότι χρειάζεται να υπάρχει μια επανεξισορρόπηση της σχέσης μεταξύ του τι θέλουν, τι χρειάζονται οι γεωργοί και τι κάνουν τα κατά τα κατά Υπουργεία Γεωργίας. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι με αυτά που κάνετε οι γεωργοί προσπαθούν κάθε μέρα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και με αυτά που κάνετε τους έχετε κάνει εχθρούς σας. Ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Συμφωνώ μεν, όμως όχι, δεν είναι εχθρός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ. Είμαι εισηγητής της γνωμοδότησης από πλευράς Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής. Έχουμε εγκρίνει την ε, έκθεσή μου και οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε και οι συστάσεις που περιέχει το κείμενο κατά τη γνώμη μου αναδεικνύουν τα εξής θέματα. Όσο γίνεται λιγότερα ζητήματα να αριθμιστούν με κατεξουσιοδότηση πράξης η βασική νομοθεσία να λύσει τα ζητήματα και να τα ρυθμίσει. Δεν θέλουμε η ΚΑΠ να διέπεται από κάτι εξουσιοδότηση πράξης. Θέλουμε τις βασικές αυτόνομες νομοθετικές πράξεις. Έχουμε βάλει σχετικέ τροπολογίε για κάποια σημεία όσον αφορά την προθεσμή του Φεβρουαρίου που θέλουν να πάει τον Απρίλιο γιατί είναι αδύνατον τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να υποβάλουν τις εκθέσεις των επιδόσεών τους τόσο γρήγορα. Είναι εκθέσεις που αφορούν την προηγούμενη χρήση. Επίσης, για τις εκθέσεις ε, να παραμείνει το ισχύον σύστημα. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο εντελεγής αυτέ οι εκθέσει όπω κάνουμε με τις εκθέσεις Περιφερειακή Πολιτική για τα ταμεία συνοχή. Τώρα, όσον αφορά το κριτήριο της ανωτέρας βίας, Θέλουμε ότι οι φυσικές καταστροφές θα πρέπει να καλύπτουν και τον θάνατο του επικεφαλής ε, της κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης. Ο θάνατος του αρχηγού της οικογένειας του ΣΥΠΗΝ είναι χειρότερος από θεομηνία, από φυσική καταστροφή για την εκμετάλλευση. Προσοχή λοιπόν σε ένα σημείο που σας είπα, μια που η έκθεση το τονίζει. Οι πληρωμές που έχουν όριο το 50% θα πρέπει μόνο τον πρώτο πυλώνα γιατί οι κύκλοι των δημοπρατήσεων ε, είναι πολύ περιορισμένες. Πολύ περιορισμένοι για αυτόν τον κλάδο. Ο κύριος Ντεκάστρο. Συμφωνώ με την Ούλρικα Μίλλερ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει τώρα να, να ε, προχωρήσουμε από το σημερινό ε, σύστημα τη συμμόρφωση προ τον νόμο σε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται ε, στι επιδόσει τη παραγωγή. Άρα αυτό άρα είναι βασικό ο δεύτερο πυλώνα και σωστά τονίζεται ότι υπάρχει ένα κίνδυνο συγχρηματοδότηση για το σύνολο τη ΚΑΠ. Και επ' αυτού εγώ αναρωτιέμαι ακριβώς ποιον αφορά αυτή η καινούργια συγχρηματοδότηση για το νέο μοντέλο. Αυτό σίγουρα δεν αφορά τους ε, γεωργούς, γιατί σίγουρα ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και τις ε, στρεβλώσεις που θα προέλθουν. Αν έχουμε επομένω ε, του κοινού κανόνε όπω με το σημερινό σύστημα, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ισότητα μεταχείρισης με κάποιον έλεγχο ετήσιο όσον αφορά την επίδοση σε βάθος χρόνο. Και πλέον η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνεται από τρίτους φορείς και όχι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως και κάποια απλούστευση θα προκύψει, αλλά αυτό δεν θα ωφελήσει τους ε, γεωργούς οι οποίοι θα πληγούν από τις ε, χρηματοοικονομικές ή δημοσιονομικές διορθώσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να σας πω κάποιες σκέψεις μου πρώτα-πρώτα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η πρικοδότηση θα πρέπει να είναι λιγότερη από ό,τι στην περίοδο 14-20. Υπό αυτό το πνεύμα κάναμε την ψηφοφορία. Το δε Brexit είπαμε ότι δεν θα πρέπει να το πληρώσει η κοινή γεωργική πολιτική. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν έχουν το κουράγιο να συζητήσουν το πολιτές δημοσιομικό πλαίσιο το Δεκέμβριο και θα μεταθέσουν την ευθύνη στους διαδόχους τους. να έχουμε κατά νου ποιοι είναι οι στόχοι μας και ποιες θα είναι οι συνέπειες του ότι κάποια πράγματα δεν θα διεκπαιρεωθούν τώρα. Αυτά να τα ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, όσον αφορά την βιολογική γεωργία και την ε, προοικοδότησή της, παρουσιάζει ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Ε, τώρα καλύπτεται η βιολογική γεωργία από τον δεύτερο πυλώνα. μπορεί κανείς να προσφέρεται να κάνει αυτή τη δραστηριότητα αλλά από την άλλη μεριά η χρηματοδότηση γίνεται με πολύ αυστηρούς κανόνες γιατί είναι πολύ πιο ακριβή αυτή η γεωργία. Δεν θα πρέπει να ασκείται αυτή η δραστηριότητα βάρος των υπολείπων μη βιολογικών γεωργών. Μην τους φέρουμε σε αντιπαράθεση αυτούς τους δύο κλάδους. Οπότε, ας προβληματιστούμε για τη χρηματοδότηση της βιολογικής παραγωγής από τους, ε, το σύνολο των Ευρωπαίων ε, ε, γεωργών. Πρέπει να αποδείξουμε ότι θέλουμε να υποστήριξουμε τη βιολογική γεωργία και όταν κάποιο ε, θέλει να γίνει βιολογικό γεωργό, να μπορεί να το κάνει. Όχι να περιμένει μέχρι να μαζέψει τα πάρει τα λεφτά. Θα πρέπει όταν έρθει η ώρα να τεθούν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί, να λύσουμε το πρόβλημα των εφαρμοστικών κανόνων και να επιλύσουμε επίση και το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Κύριε Στάση, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την κυρία Μούλη για την παρουσίαση της εργασίας ως τώρα. Να περιοριστώ σε κάποια θέματα σε ό,τι αφορά την κρίση στις άλλες χώρες αναφέρθηκαν τα διάφορα ζητήματα. Το θέμα είναι πώς θα οργανωθεί ο έλεγχος, γιατί ε, η αλλαγή των κανόνων ε, πιστεύω σήμερα δεν έχει είναι σκόπιμη το θέμα είναι πώ θα αντιμετωπίσουμε την κριτική στην πολιτική γεωργία. Σε ένα παράδειγμα, το είπε ο Ιρλανδό συνάδελφο, υποχρεωθήκαμε να καταθέσουμε ένα πενταετέ σχέδιο σε ό,τι αφορά τον τομέα των ε, λουλουδιών. Πρώτο χρόνο λοιπόν, δεύτερο χρόνο, ε, μειώθηκε η παραγωγή λουλουδιών την τέταρτο χρόνο ουσιαστικά μείωσε η ίδια η φύση την παραγωγή. Πέτυχα χάρα για το στόχο μου ή όχι. Παρ' αυτά ε, ήταν σωστοί οι κανόνες και η φύση πολύ απλά δεν συνεργάστηκε. Θα πρέπει να ορίσουμε το στόχο λοιπόν αυτόν αν ε, το τεταρτο ο 5 ακόμα δεν έχουμε πετύχει τον ε, στόχο μας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε ρεαλιστικούς στόχους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους στόχους. Είναι μη ρεαλιστικό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στο τρέχον σύστημα. Πληρώνουμε τους ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο όταν πετυχαίνουν τους στόχους τους. Το κατά πόσο λοιπόν έχουν επιτευχθεί η στόχη, πιστεύω ότι δεν μπορεί να έχει επίπτωση στο κατά πόσο θα πληρώνουν τα χρήματα αυτά. Α παραμείνουμε λοιπόν στο τρέχον σύστημα, γιατί κατά τα άλλα νομίζω ότι θα βλάψουμε και μόνο το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Μπούντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. και θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. κάποιε ερωτήσει για την απλοποίηση. Φυσικά θέλουμε όλοι να πετύχουμε μια απλοποίηση, πραγματική απλοποίηση. Και θα πρέπει να επιμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκαθαριστεί ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις προκειμένου τα κράτη-μέλη να μην έχουν την δυνατότητα να εισαγάγουν νέα αρεσιμότητα στο επίπεδο αυτό. Στη συνέχεια έχουμε το θέμα της απόδοσης, performance. Αγαπητοί συνάδελφοι, ό,τι και να λέμε, είτε λέμε απόδοση, είτε χρησιμοποιούμε κάποιον άλλον όρο, το θέμα είναι οι μηχανισμοί αυτοί που είναι απαραίτητοι γιατί μιλάμε για δικαιούχους, δικαιούχους επιδοτήσεων που ασχολούνται με τη Γεωργία. Κάποια κρατημέλη, μεταξύ των οποίων και η Ρουμανία, χαρακτηρίζονται από μεγάλη κερδοσκοπία σε ό,τι αφορά τις τιμές των ε, προϊόντων. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, αγροτικοί τομείς που ωφελούνται από τις επιδοτήσεις χωρίς όμως να παράγουν τα αντίστοιχα. Άρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει παραγωγή Υπάρχει παραγωγή προϊόντων που αξίζουν να επιδοτούνται. Φυσικά λοιπόν μπορώ να πω διάφορα για το θέμα αυτό. Ο κύριος Ντες για παράδειγμα ανέφερε τον τομέα των ανθέων σε ό,τι αφορά την πενταετία αυτή περίοδο που είχε προβλεφθεί η καλλιέργειά του κτλ. Το θέμα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το ακολουθήσουμε πέντε χρόνια και θα πρέπει να υπάρχει και έλεγχος στο χρονικό αυτό διάστημα. Ιδάλλως θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου τα χρήματα τελικά θα πηγαίνουν σε άτομα τα οποία δεν ασχολούνται καν με τη γεωργία. Ένα τελευταίο στοιχείο τώρα, επιτρέψτε μου να αναφέρω. Η γεωργοί. Οι οποίοι περνούν από έλεγχο. Θα πρέπει να έχουν και ανάλογες χρηματικές δυνατότητες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια ο κύριος Γιάρ. Τέσσερα-πέντε σημεία έχω σημειώσει. Το πρώτο λοιπόν θέμα, όπως είπε σωστά η συγγήτρια, θα πρέπει να κοιτάξουμε να υπάρχει συνοχή μεταξύ των εκθέσεων. Δεύτερο μεγάλο ζήτημα για μένα. Από γραφειοκρατικοποίηση. Αυτό μας υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να φτάσει και μέχρι τη Γεωργία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην ξεχάσουμε τους γεωργούς στο όλο παιχνίδι. Φυσικά και αλλού να υπάρχει μείωση τη γραφειοκρατίας, αλλά και στη γεωργία. Και να μην καταλήξουμε να ελέγχουμε τον έλεγχο. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του λάθους και της απάτης. Αυτό κάπου μπορούμε να αναφέρουμε. Τρίτον, τα περιβαλλοντικά προγράμματα. Τα συζητήσαμε επισταμένως στη διαδικασία του greening. Τα περιβαλλοντικά αυτά προγράμματα έχουν νόημα μόνο εφόσον υπάρχει μια πολιτική εφαρμογή. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε μετά από λίγο καιρό. Γι' αυτό λοιπόν είμαι κατά των ελέγχων αυτών. Τέταρτο, η αρχή ε, της αναφοράς ε, στην ε, επίδοση και όχι στους κανόνες. Ωραίο ακούγεται αυτό με την επίδοση και την απόδοση, αλλά νομίζω ότι στην πράξη αυτό θα δημιουργήσει πιο πολλά προβλήματα από ότι θα λύσει. Να πω ένα παράδειγμα πέρα από αυτό που είπε ο συνάδελφο, γιατί είμαι κατά τον έλεγχο της απόδοσης Το πρόγραμμα για την συσταξονία ε, το είχαμε κάνει αυτό για πολύ πολύτιμα, πολύτιμες καλλιέργειες. Μπορούμε να κοιτάξουμε αν καλλιεργείται ή κατά πόσον αναπτύσσεται. Ωραία ακούγεται αυτό στην θεωρία, αλλά γενικά δημιουργεί πιο πολλά προβλήματα από τη λύνει. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι ενδεχομένως και να πρέπει να συζητήσουμε σε μετέπειτα χρονική στιγμή αυτό το ζήτημα της αλλαγής του συστήματος σε ένα σύστημα απόδοσης. Επίσης, είμαι υπέρ του να είναι όσο πιο περιορισμένες γίνεται η πράξη κατά εξουσιοδότηση. Όχι επειδή δεν εμπιστεύομαι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση ακόμα, και το λέω αυτό, ακόμα και την ε, βούληση της Επιτροπής μας να ε, προωθήσει. Αλλά πιστεύω παρόλα αυτά θα πρέπει να είναι όσο πιο λίγες γίνονται αυτές οι πράξεις κατεξιδότηση. Ο κύριος Χόσλινγκ, ευχαριστώ. Είπε μια πρόταση στην αρχή η κυρία Μιούλερ, την οποία θα ήθελα να μου την εξηγήσει, ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει. Μα τι δεν θα λειτουργήσει. Αυτά που υπεβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ε, πρόταση ή το όλο σύστημα, γιατί νομίζω ότι επισερχόμαστε σε πολλές λεπτομέρειες. Όλοι έχουν ερωτήσεις, γιατί προφανώς ε, καμία από τις ε, ερωτήσεις δεν έχει απαντηθεί επαρκώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, αλλά πολύ λίγα συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς θα διαμορφωθεί αυτό το νέο σύστημα και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και εκεί αποτυγχάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό λοιπόν καθόμαστε και το συζητάμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ως κοινοβούλιο πώς θα αποδώσουμε, θα ε, πετύχουμε αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς λεπτομέρειες. Ε? Ωραία, να αλλάξει το σύστημα. Το, να θέλουμε να αλλάξει, δεν θέλουμε να αλλάξει. Αν θέλουμε να αλλάξει, προφανώ υπάρχουν και λόγοι για του οποίου μπορεί να θέλουμε να αλλάξει το σύστημα, αλλά να ξέρουμε τελικά τι αποτέλεσμα θέλουμε να πετύχουμε. Και εδώ δεν έχω λάβει ακόμα αποφα... Ε, απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θέλουμε να πετύχουμε. Τι θα κάνουμε, θα πούμε δηλαδή στα κρατημέλη, αποφασιστείτε εσείς τι αποτέλεσμα θέλετε να πετύχετε. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πολλά διαφορετικά αποτελέσματα τα οποία θα αποφασιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όλα αυτά θα τα ελέγξουμε και θα τα ονομάσουμε ένα σύστημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Και αυτή η επανεθνικοποίηση τη πολιτική, τη γεωργική πολιτική είναι τεράστιο σφάλμα. Αν συνεργαστούμε σε αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να θάψουμε και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να πω αυτό ξεκάθαρα. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει αυτό. Κατά δεύτερον, γραφειοκρατία. Εδώ το θέμα ήταν μείωση γραφειοκρατία. Μα δεν είδα πουθενά να το πετυχαίνουμε αυτό. Και προφανώ υπάρχουν και πολλοί δικαιολογημένοι φόβοι ότι τα κράτη-μέλη τελικά θα καταλήξουν να διαμορφώσουν τα συστήματα με πιο περίπλοκο τρόπο, όχι να τα απλοποιήσουν, ε, αλλά να τα περιπλέξουν. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να κοιτάξουμε το κείμενο άρθρο προς άνθρωπο γίνεται σε άλλα αναμορφωτικά ε, κείμενα, αλλά να δούμε καταρχά ω σύστημα, ω αρχή μπορεί να λειτουργήσει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαντλήθηκε ο κατάλογος ομιλητών. Τώρα. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ, κύριε Βόρκουμεν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Προσπάθησα να ακούσω πολύ προσεκτικά τις παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών. Αυτό που θέλω να τονίσω έχοντας ακούσει τις επικρίσεις σας ναι, να σας πω τι ακριβώς θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το νέο οριζόντιο αυτό κανονισμό και με το σύστημα επιδόσεων. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις επικρίσεις που έχουν ακουστεί επίση από αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το διοικητικό άχθος του τρέχοντος συστήματος συμμόρφωσης με πολύ λεπτομερείς κανόνες. Και θέλαμε επίση να ενισχύσουμε και τα αποτελέσματα, την αξιολόγηση βάση αποτελεσμάτων. Εξού και είναι αυτή η πρόταση. Όπως είπατε πολλοί από εσά, περνάμε από την ε, συνολική συμμόρφωση στην ατομική επίδοση που συμπληρώνεται με τις επιδόσεις των χωρών μελών. Κάποιοι από εσά ε, είπαν εμείς δεν θέλουμε την ε, επίδοση στο επίπεδο του Γεωργού. Αλλά δεν είναι αυτό που προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζουμε συγκεκριμένους κανόνες επιλεξιμότητας για τον κάθε δικαιούχο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα γίνονται βάση των επιδόσεων. Πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση προς τους κανόνες. Λέμε ότι θέλουμε να επικεντρωθούμε στις επιδόσεις, αλλά όχι ατομικά του κάθε γεωργού, γιατί και ο κ. Φλάνεγαν το είπε, δεν είναι το τι κάνει ο κάθε δικαιούχος που μετράει σαν αποτέλεσμα, αλλά το τι κάνει συνολικά σε μια χώρα το σύνολο των γεωργών. Έτσι υπολογίζουμε τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Πολλοί επίση είπαν ότι υπάρχουν γεωργοί που τηρούν τους κανόνες, αλλά κανόνες δεν έχουν νόημα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν νόημα. Θέλουμε επιδόσεις βάσει των ευρωπαϊκών στόχων και ζητούμε από τις χώρες μέλη να συμμορφωθούν, να θέσουν στόχους για αυτές τις ε, επιδόσεις, για αυτά τα αποτελέσματα και μετά οι χώρες μέλη να μας πούνε τι κανόνες πρέπει να τεθούν για τον κάθε δικαιούχο, τι είναι το ελάχιστο που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε τα αποτελέσματα χωρίς να έχουμε τους ίδιους κανόνες για όλους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια παραδείγματα για τους, ε, τις τοποθεσίες που είναι ευαίσθητες οικολογικά, που είναι στην περιφέρεια, στα παράκτια κτλ. Λένε οι χώρες ποιο μπορεί να είναι το όριο, τι εξαιρέσεις μπορεί να υπάρχουν. Οπότε αρχίζουμε να ε, καταρτούμε και κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ έχω ταξιδέψει σε όλες τις χώρες μέλη και κοίταξα να δω πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, ε, οι φράχτες ας πούμε στις καλλιέργειες, στην Ιρλανδία ή στην Πολωνία, στο γεωργικό τοπίο, στην Ήπεθρο είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Οπότε τι λέμε σε αυτή την πρόταση είναι ότι θα θέλαμε να μπορούσαμε να έχουμε χώρους ε, οικολογικούς, να υπάρχουν ε, επιδοτήσεις για την ε, διατήρηση αυτών των χώρων, αλλά αλλού δεν υπάρχουν καθόλου. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διευθετήσουμε. Ο καλύτερος τρόπος είναι να αφήσουμε τις χώρες μέλη να αποφασίσουν για αυτές τι σημαίνει ακριβώς αυτός ο φράχτης από φυτά. Και ανάλογα να αποφασίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα ζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε λεπτομερείς κανόνες για τους δικαιούχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το επίπεδο επιδόσεων θα ήταν το δεύτερο επίπεδο και θα είχαμε ακόμα περισσότερο διοικητικό άξονα από ό,τι έχουμε σήμερα. Ε, καταλαβαίνω ότι η κυρία Μίλλερ μιλάει και για τη μεταβατική περίοδο. Εδώ έχω να πω ότι εμείς δεν λέμε ότι απομακρυνόμαστε πλήρως από την συμμόρφωση και πηγαίνουμε 100% στις επιδόσεις. Όχι, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά συστήματα ελέγχων στις χώρες μέλη που λειτουργούν και για να μην δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες δυσκολίες, λέμε στις χώρες μέλη, συνεχίστε με ό,τι λειτουργεί καλά στις χώρες σας. Είτε έχετε υπηρεσίες πληρωμών, είτε έχετε συστήματα εντοπισμού κτλ. Όλα αυτά τα δεχόμαστε με την πρόταση της Επιτροπής, ότι λειτουργεί καλά τώρα και που δεν θα αποτελεί διοικητικό άχθος για τη χώρα μέλη, θα συνεχί... μέλος θα συνεχίσει να υπάρχει. Όσον αφορά τους δικαιούχους και ποια θα είναι για αυτούς η απλοποίηση. Όπως είπα και πριν, η πρόθεσή μας και αυτό που προβλέπετε είναι να μην υπάρχουν κανόνες σε επίπεδο δικαιούχων που να μην έχουν νόημα για το συγκεκριμένο δικαιούχο. Η χώρα μέλος δηλαδή αποκτά την ευελιξία να μπορεί να καθορίσει εκείνη τους κανόνες στην ίδια τη χώρα ή σε κάποια περιφέρεια που να έχει νόημα για τη συγκεκριμένη περιφέρεια, για τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό είναι το νέο μας μοντέλο. Και σας ακούω να λέτε πολύ ότι δεν θα λειτουργήσει. Και αναφερθήκατε στην ημερομηνία της 15ης Φεβρουαρίου. Τι κάνουν οι χώρες μέλη τώρα. Μας ε, κάνουν συγκεκριμένες δηλώσεις για την κανονικότητα και νομιμότητα και μας δίνουν ε, στοιχεία για όλες τις πληρωμές που έχουν γίνει ατομικά για τον κάθε δικαιούχο. Δεν θα φτάσουν μέχρι τον τελευταίο δικαιούχο. Αυτό λοιπόν που ζητάμε εμείς για τις 15 Φεβρουαρίου δεν είναι ατομικά τα αποτελέσματα, αλλά συνολικά τα αποτελέσματα. Αυτό θέλουμε. Και θα βεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία από το όργανο πιστοποίησης, που τώρα όμως πιστοποιούν την κανονικότητα και την νομιμότητα των δαπάνων για κάθε δικαιούχο. Είναι κάτι διαφορετικό δηλαδή που θα μας στείλουν έχει να κάνει με την επιλεξιμότητα των δαπανών. Αλλά εμείς δεν θα ζητάμε το λεπτομερές. Είναι δύσκολο. Γιατί αν λέτε ότι θα είναι πολύ άχθος για τις χώρες μέλη να κάνουν τέτοιες εκθέσεις με συνολικά τα ποσά στο μέλλον, ε τότε τι θα πούμε για αυτό που κάνουν σήμερα, που φτάνουν στον τελευταίο δικαιούχο. Και απλώς οι οργανισμοί πιστοποίησης θα πιστοποιούν τα ποσά που θα δίνουν οι χώρες μέλη, ο αριθμό των ε, εκταρίων για παράδειγμα, θα πιστοποιείται ή των προγραμμάτων για εξυγχρονισμό των ε, καλλιρών και της παραγωγής. Τώρα αυτά τα πράγματα δεν πιστοποιούνται, στο μέλλον θα πιστοποιούνται από το όργανο πιστοποίησης, που όμως δεν θα εξετάζουν ατομικά την κάθε περίπτωση για να δούνε τις δαπάνες και την ομότητα και την κανονικότητα της κάθε δαπάνης. Προσπαθούμε λοιπόν να πούμε ότι θέλουμε να ελαφρύνουμε από το διοικητικό άκθος και να έχουμε μόνο κανόνες που έχουν νόημα για να πετυχαίνουμε τους στόχους και συγχρόνως να βελτιώσουμε τις επιδόσεις. Αυτό λέει το νέο μοντέλο και αυτό προτείνει και ο οριζόντιος κανονισμός. Βέβαια, με ενδιαφέρον διαβάσαμε όλες τις τροπολογίες που έχουν ε, κατατεθεί για τον οριζόντιο κανονισμό. Πολλές ανησυχίες ισχύουν, αλλά πάρα πολλές το είπε και ο Επίτροπος ότι μπορούν κάλλιστα να καθησυχαστούν. Και γι' αυτό είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να βρούμε συμβασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχει μισή ώρα ο κύριο Φιλάναγκελ τώρα. Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό μου Πρόεδρε. Μα είπατε για τους φράχτες από τους θάμνους, από φυτά, τη συντήρησή τους και η κυρία Μαγκίνε το έχει αναδείξει επανειλημμένα, δηλαδή να πληρώνονται κάποιοι για να τοποθετούν αυτούς τους φράχτες. Δηλαδή έχουν προϋπάρξει αλλά θα πρέπει κάπως να εξασφαλιστεί το ότι δεν θα τα ξεριζώνουν επίτηδες για να παίρνουν τα λεφτά. Θα πληρώνουν τη συντηρησή τους ή όχι. Πώς θα γίνεται η φύτευσή τους και από την άλλη μεριά. Πώς θα παρακάμψουμε τον κίνδυνο ε, της εκρίζωσης. Μπορείτε να απαντήσετε, κυρία Μαγκίνας. Όχι, η Επιτροπή, όχι, όχι. Ε, δεν είναι δυνατόν να κάτσουμε να νομοθετήσουμε για το πόσο ε, θα είναι αυτή η φράχτες, ούτε θα είναι η απόσταση μεταξύ τους. Ναι, ε, να, να υπάρξει κάποιο είδου επιδότηση ε, υπέρ της βιοπικιλότητας. Να δούμε πώς μπορεί ο καθένας να βοηθήσει για να πετύχουμε αυτό μας τον στόχο. Να δούμε και τα κράτη-μέλη. Τι είναι διατεθειμένα να πληρώσουν για την επιτυχία αυτών των στόχων. Αυτή είναι η πρότασή μας. Κύριε Μαγίνες, όχι δεν ήθελα να το λόγο, αλλά ξέρετε πολύ συχνά ασχολούμαι με τους ε, φράχτες και με το κατά πόσον θα μπουν εκεί που δεν πρέπει τα πρόβατα. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε μια πολύ άρτια απάντηση. Έχουμε την έκθεση των κρατών μελών που θα είναι απλούστερη της τώρα ε, συντασσόμενης. Και θα πρέπει να δούμε όμως να μην ζητάει και περισσότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον κάθε Γιωργό Το κράτος, το κράτος μη ζητάει περισσότερο από το. Και αν δεν υπάρχει συνεννόηση, πώς θα υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία στις σχέσεις Γιωργού και ε, κράτους. Θα ήθελα αυτό να μου σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον επόμενο στην Επιτροπή και τα κρατημέλη έχουν πει ότι παρέχουμε πολλούς λεπτομερείς κανόνες που δεν ωφελούν όλους τους δικαιούχους. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να γίνει στενή συνεργασία με τα κρατη και τα κρατη να ξέρουν ακριβώς τι κανόνες χρειάζεται να συνεχίσουν να εφαρμόσουν. Και τι θα ισχύει σε κάθε χώρα, σε κάθε περιφέρεια χώρας. Σήμερα θα συζητήσουμε κι άλλο κανονισμό και θα τα ξαναπούμε. Αλλά όταν έρθει η ώρα τη έγκρισης του στρατηγικού προγράμματος, τότε θα το ξαναδούμε εμεί στην Επιτροπή. Θα εγκρίνει αυτό το στατικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Επιτροπή οπότε ταυτόχρονα θα δούμε τις απλουστεύσεις που θα περιέχει αυτό το πρόγραμμα και αυτό αφορά και τον κανονισμό αλλά όχι τον κανονισμό για στρατηγικό πρόγραμμα αλλά όχι τον κανονισμό τον οριζόντιο ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ανταλλαγή αυτή απόψεων και για τις παρατηρήσεις που κάναν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε με σαφήνεια το πόσο αμφιλεγόμενη είναι η συζήτηση, πόσα ζητήματα είναι εκκρεμή και πόσε ερωτήσει ακόμα παραμένουν εκκρεμή. Νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ότι ω εισηγήτρια θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό με όλη την ομάδα και να κοιτάξουμε καταρχά προ τα πού θέλουμε να οδεύσουμε, πού θέλουμε να καταλήξουμε και να κάνουμε συμβαστικέ τροπολογίε προ την κατεύθυνση αυτή. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Επίση, ε, Πρόεδρε, μα ζητήσατε να πούμε τι γίνεται με του δείκτε σε ό,τι αφορά το σεμινάριο τη ΑΛΔΕ. 6 του μηνό στην ε, αίθουσα Γιάν έχουμε από αγγλικά, στα αγγλικά, γερμανικά και ε, γαλλικά διερμηνία θα λάβετε και τις επίσημες προσκλήσεις στο σεμινάριο λοιπόν αυτό της Άλντα για τους δείκτες. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας για τον οριζόντιο αυτοκανονισμό προκειμένου να προχωρήσουμε. Δεν θα είναι εύκολο να τους ικανοποιήσουμε όλους, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ επικοδομητική. και πραγματικά θεωρούμε ότι ενημερωθήκαμε σωστά για το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμφωνήσει και αυτή μαζί μας. για την ε, απλοποίηση, την απλούσταυση. Αυτό θέλουμε να είναι το αποτέλεσμα του κανονισμού αυτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Φεράνς Γκαρσία έχει καταφτάσει. Καλώς ορίσατε. Και έτσι λοιπόν, χωρίς να καθυστερήσουμε, να μας δώσω το λόγο Αναμένουμε ακόμα την γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Θα είναι πολύ σημαντική βάση του άρθρου 54. Αναμένουμε και άλλες γνωμοδοτήσεις, αλλά προτού α, ακούσουμε τις τοποθετήσεις αυτές, να δώσουμε το λόγο στην εισηγητρία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτές τις εβδομάδες δουλέψαμε πολύ σκληρά. Ολόκληρη η ομάδα μου και οι συνεργάτες μου και θέλω να τους ευχαριστήσω. Μην το ξεχάσω μετά. Ευχαριστώ και το προσωπικό της γραμματείας και της πολιτικής μου ομάδας που συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά μαζί μας. Αυτές τις εβδομάδες λοιπόν είχαμε 13 τεχνικές συναντήσεις Κάτι το οποίο σας δίνει μια ιδέα για το με τι ρυθμό εργαστήκαμε για το θέμα αυτό και είχαμε και τρεις συναντήσεις σκιωδών εισηγητών. Έχουν ετοιμαστεί άλλες 15 τεχνικές συναντήσεις και άλλες τρεις με τους σκιώδες εισηγητές. Γιατί δεδομένη της ημερομηνία της ψηφοφορίας πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να αφήσουμε ανοιχτέ όλε τις δυνατότητες. Όλοι είναι ανοιχτά λοιπόν από πλευρά των πολιτικών ομάδων και από τους πράσινους και από τους σοσιαλιστές και από την ΚΟΕ. Από την αρχή το μήνυμα που είχαμε ότι αν δεν υπάρχει ένα τελικό αποτέλεσμα όλα παραμένουν ανοιχτά. Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί, δεν έχουν αποφασιστεί όλα δηλαδή. Επιφυλάζονται πώς θα ψηφίσουν, αν θα ψηφίσουν υπέρ ή κατά, ανάλογα με την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Όλα λοιπόν είναι ανοιχτά. Έχουμε όμως προχωρήσει. Ουσιαστικά έχουμε προχωρήσει. Επικεντρώσαμε τη διαπραγμάτευση από την αρχή σε ένα θέμα που είναι ο πρώτος πυλώνας της κοινή γεωργικής πολιτικής. Γενικοί στόχοι, γενικές γραμμές, δηλαδή και πρώτος πυλώνας της κοινή γεωργικής πολιτικής. Όσον αφορά τους στόχους, πρέπει να σας πω ότι έχουμε γεμίσει με στόχους. Έχουμε συμπληρώσει δηλαδή τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πιο πλήρης η στόχη δηλαδή με την ε, βοήθεια των πολιτικών ομάδων. Υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό και αυτό είναι ο ρόλος της γυναίκας στην κοινή γεωργική πολιτική. Υπήρξαν τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση που τις ε, δεχτήκαμε. Όσον αφορά τους δείκτες τώρα. Και εδώ η συζήτηση παραμένει ανοιχτή. Γενικά μιλώντας το ΕΛΚ, οι φιλελεύθεροι, το ECR, στηρίζουν την δικιά μας γραμμή, αλλά οι σοσιαλιστές θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξουν στόχοι για τους δείκτες επιπτώσεων. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι μια δυσκολία, δεν γίνεται. Αλλά οι σοσιαλιστές επιμένουν. Όσον αφορά τους ορισμούς, τους μεγάλους ορισμούς, εδώ πρέπει να σας πω ότι τι σημαίνει αυθεντικός γεωργός. Αυτό είναι το βασικό που μας δημιουργεί η δυσκολία δεν έχουμε προχωρήσει πολύ στους ορισμούς για το ότι είναι πραγματικός Γιώργος. Ελπίζω όμως να καταφέρουμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά τώρα και για τα, τους μόνιμους βοσκοτόπους. Εδώ οι γεωργοί εντυπωσιάζονται από τα πέντε χρόνια προκειμένου να είναι μόνιμα τα βοσκοτόπια. Είναι μια καινοτομία αυτή, είναι μια δυσκολία που πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε μεταξύ μας. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες θέσεις ως ομάδα, μας στηρίζουν και κάποιες άλλες πολιτικές ομάδες. Θα συνεχίσουμε και εδώ ε, τη δουλειά. Τώρα για τους νέους γεωργούς, εδώ έχουμε συστήσει πάρα πολύ, δεν υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες εδώ. Και για αυτούς που είναι νέοι γεωργοί, όχι στην ηλικία, αλλά νέοι στο επάγγελμα του Γεωργού, ε, πιστεύουμε ότι και εδώ μπορούμε να έχουμε συμφωνία. Στους γενικούς στόχους επιμένει για την εξωτερική σύγκληση η σοσιαλιστική ομάδα. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι στα εθνικά σχέδια, πρέπει να είναι κάτι εξωτερικό. Και μετά περνάμε στην αιρεσιμότητα. Τα σημεία 11, 12 και το παράρτημα 13. Στα άρθρα 11, 12 και το παράρτημα 13 έχουμε έναν από τους βασικούς πυλώνες σχεδιασμού των στρατηγικών σχεδίων. Η δικιά μας ιδέα βρίσκει σύμφωνος πολλούς στην Επιτροπή Γεωργίας ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ενιαία αντιμετώπιση της κοινή γεωργικής πολιτικής όσον αφορά αυτό το θέμα της αιρεσιμότητας. Υπάρχει λίγο πολύ μια συμφωνία, αλλά παραμένουν κάποιες διαφορές για το κατά πόσο τα δικαιώματα των εργαζομένων και το κοινωνικό σκέλος θα πρέπει να διακανονίζεται στο άρθρο 11 ή όχι. ΕΛΚ, ΑΛΔΕ και ΙΣΙΑΡ δεν συμφωνούμε. Οι σοσιαλιστές όμως το προτείνουν και επιμένουν με τη στήριξη των Πρασίνων και της ΓΚΟΕ. Όσον αφορά το άρθρο 12. Είναι εδώ η Σοφία Ριπέιρο και οι άλλοι συνάδελφοι από τις ε, απόμακρες περιοχές. Εδώ δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Όταν μιλάμε τώρα για τα ισοδύναμα στις καλλιέργειες, εδώ είναι κάπως πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά οι περισσότερες πολιτικές ομάδες στηρίζουν τον ορισμό Στο παράρτημα τώρα. Εδώ υπάρχει μια γενική συμφωνία θα έλεγα. Και κυρίως εδώ θίγεται κάτι πολύ ενδιαφέρον για την κοινή γνώμη, για την κτηνοτροφία. Πρέπει να σας πω ότι εδώ δεν είναι τόσο το θέμα της υποχρέωσης του εντοπισμού των ε, ζώων, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα και να επιβαρυνθούν οικονομικά οι αγρότες. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για αυτό το θέμα, γιατί εμείς στο ΕΛΚ θεωρούμε ότι αυτή η τιμωρία κατά κάποιο τρόπο, πώς αλλιώς να το πω, σε βάρος των αγροτών για κάτι που δεν μπορούν να αποφύγουν, πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικό. Εντάξει να υπάρχει έλεγχος ε, των ε, κοπαδιών, αλλά όχι και να τιμωρούμε τους αγρότες, οι οποίοι δεν μπορεί 24 ώρες στις 24 να είναι δίπλα και να είναι σίγουροι ότι το ενότιο στα ζώα τους βρίσκεται στη θέση του και δεν έχει φύγει. Και εμείς χάνουμε καμιά φορά κανένα σκουλαρίκι, κανένα δαχτυλίδι κανένα βραχιόλι, φανταστείτε τι γίνεται με τα ζώα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να συζητάμε και αυτό το θέμα. Στην υπόλοιπα έχουμε προχωρήσει πολύ. Έρχομαι τώρα για τη στήριξη των ε, καλλιεργιών. Αυτό που είναι ενδιαφέρον εδώ είναι ότι πολλοί εξέφρασαν ανησυχίες για αυτοκτονίες, για αρρώστες, κατάθλιψη των ε, αγροτών συχνά. Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει κάποια λύση ώστε να ληφθεί υπόψη αυτή η στήριξη. Να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή και την υγεία τόσο την σωματική όσο και την ψυχική των αγροτών και των οικογένειών τους στην Ήπεθρο. Ένα άλλο πολεμικό ζήτημα που πολύ αναφέρεται και στον τύπο εμένα Πάντα με ρωτάνε Μιλάμε για 50.000 το ανώτατο όριο, το κάπινγκ. Δεν θα εφαρμόζεται εάν η χώρα μέλος αποφασίσει το 5% να το δώσει αναδιαναμητικά. Αυτός είναι και ο στόχος του κάπινγκ. Εδώ είμαστε πολύ διχασμένοι μεταξύ μας. Δεν βλέπω ακόμα τι κατεύθυνση θα πρέπει να πάρουμε. Οι πράσινοι, οι γκου, οι σοσιαλιστές είναι σαφώς κατά. Το ECR, οι φιλελεύθεροι και το ΕΛΚ ακολουθούμε διαφορετική γραμμή. Θα δούμε αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι. Θα ήταν ενδιαφέρον να πετύχουμε μια πλειοψηφία να μας στηρίξει. Πάντως οι ιδέες αυτές, του να λάβουμε υπόψη μας τις αμοιβέ όταν πρόκειται για δηλωμένη βέβαια εργασία, το δέχονται όλοι. Αυτό που δεν δέχονται είναι το εισαδύναμο του κόστους μιας εργασίας που δεν είναι δηλωμένη γιατί στις οικογένειες, στις εκμεταλλεύσεις συμβαίνει αυτό. Δεν το θέλουν οι πολιτικές ομάδες και ούτε θέλουν να λάβουμε υπόψη μας και τις υπηρεσίες στις κτηνοτροφικές ε, μονάδες. Έχουμε αποσύρει μια πρόταση συμφωνίας για τις ελάχιστες απαιτήσει για τις άμεσες ενισχύσεις. Γιατί δεν υπήρξε στήριξη ούτε από τις πολιτικές ομάδες, ούτε τεχνικά, ούτε από τους σκιώδεις εισηγητές. Από τις 40 τόσους συμβιβασμούς, λοιπόν, αποσύρθηκε αυτό. Τώρα η συζήτηση παραμένει ανοιχτή για τη στήριξη ανά εκτάριο. Πρόκειται για το άρθρο 18. Υπάρχει λίγο πολύ μια συμφωνία που λέει ότι οι αεροκατοικημένες περιοχές με αδυναμίες θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη όλος ιδιαίτερος από τις χώρες μέλη. Επίσης να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός παράγοντας και ο αγρονομικός, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για μια πρόταση που πιστεύουμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα για χώρες όπως είναι η Γαλλία ή η Ισπανία, όπου δίνεται δυνατότητα στη χώρα μέλος να περιορίσει τον αριθμό των ε, εκταρίων που θα δικαιούνται πληρωμέ. Στην τελευταία συνάντηση σκιωδών συζητήσαμε με την κυρία Νόχελ για αυτό το σημείο. Δεν βρήκαμε λύση. Και για την κυρία Νόχελ, μια που είναι σκιώδη από τους σοσιαλιστές, πρότεινε η κατανομή αυτή να λάβει υπόψη τη συνεισφορά στο δημόσιο και έκανε μια πρόταση για το πώς το κάνουμε. Μια που μιλάμε για δημόσιο αγαθό, μια που υπάρχουν ε, περιφέρειες που προσφέρουν περισσότερα στο κράτος από άλλες, δεν χρειάζεται εδώ να δώσουμε παραδείγματα, τότε δώσαμε, πρέπει να βρούμε τρόπο να μετρήσουμε την προσφορά της μιας ή της άλλης περιφέρειας στο κράτος για να υπάρχει διαφοροποίηση. Και η διαφοροποίηση πρέπει να είναι περισσότερο στο τι μέθοδο χρησιμοποιεί ο αγρότης. Χρησιμοποιεί μεθόδους που προστατεύουν το περιβάλλον ή προσφέρουν περισσότερα στο δημόσιο. Και αυτό ανάλογα με τον παραγωγό, όχι ανάλογα με την περιφέρεια. Και για τον περιορισμό του ρυθμού των εκταρίων είναι σημαντικό για να περιορίσουμε τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων στη χώρα μου, αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήταν άσχημα τα πράγματα για τους γεωργούς. Νομίζω ότι ήταν καλό και είναι μια κόκκινη γραμμή για μας. Δικαιώματα πληρωμών. Τι ημερομηνία πρέπει να βάλουμε, ανάλογα με το πότε θα αρχίσει να ισχύει η μεταρρύθμιση. Συμβουλευόμαστε την νομική υπηρεσία. Συζήτηση που πρέπει να γίνει στο μέλλον είναι νέοι Γεωργοί. Όλοι θέλουμε να τους στηρίξουμε. Αλλά υπάρχουν διαφορές σημαντικές. Να λάβει κανείς υπόψη του τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Οι διαφορές είναι πράγματι μεγάλες. Οι νέοι αγρότες πρέπει να τύχουν της προσοχής μας. να βάλουμε κάποιες μεταβλητές στο σημερινό σύστημα για να βελτιωθεί. Παραμένει ανοιχτό και το θέμα της στήριξης για τη βιωσιμότητα. Και εκρεμεί επίσης και η συζήτηση των πληρωμών στους νέους γεωργούς. από τις 15 που έχουμε προτείνει συναντήσεις τεχνικές και άλλες τρεις με τους σκιώδεις, θα συνεχίσουμε ακριβώς αυτά τα θέματα που παραμένουν σε κρεμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τρία λεπτά για τους σκιώδεις ηγητές. Κύριε Νόχλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ράντ Καρσία. Και ναι, όντω, είναι μάλλον η φύση του θέματο ότι υπάρχουν διαφορετικέ ε, εκτιμήσει. Σα άκουσα με προσοχή και έπρεπε να προσπαθήσω να μην γνέφω συνέχεια καταχαρτικά, γιατί νομίζω ότι όλα τα περιγράφονται σωστά και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει με πάσα ειλικρίνεια να το πούμε αυτό και στο Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή, ότι δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Καταλαβαίνω ότι όλοι είναι πρόθυμοι, όλοι δουλεύουν σκληρά, όλοι έρχονται καλά προετοιμασμένοι στις συνεδριάσεις. Δεν είναι λοιπόν θέμα στήλα, δεν μας ε, χωρίζει αυτό. Όχι, το περιεχόμενο μας ε, χωρίζει. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Να ξεκινήσω με τα θέματα του δεσμευτικού χαρακτήρα κάποια ζητήματα θα πρέπει να, ρυθμούν, να ρυθμιστούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση με δεσμευτικό τρόπο. Ποια όμω και ποια θα πρέπει να μπαίνουν σε επίπεδο εθνικών κρατών μελών σε εθελούσιο χαρακτήρα. Χρειάζεται ένα στενό, καλό πλαίσιο. Το παλιό σύστημα ήταν καλύτερο, αλλά Πολλοί διάφοροι λένε, και εσείς κυρία Συγητρία ότι α, όχι, να μην είναι όλα αυτά δεσμευτικά. Όλες αυτές οι μεταβλητές να ρυθμίζονται από τα κράτη-μέλη. Άρα σε θέματα δεσμευτικού χαρακτήρα διαφέρουμε παρασάγκα. σε ό,τι αφορά το κάπινγκ. Δεν έχουμε κανένα σχέδιο για το τι θα κάνουμε ε, με τις ε, δυνάμεις εργασία, με το εργατικό δυναμικό. Κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να έρθουν οι μισθοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι πιστεύουν ότι να συμπεριθούν διαφορετικά στους εργαζόμενους. Να σας πω ότι για τους ε, ε, σοσιαλδημοκράτες δεν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο γιατί δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί να υποκρινόμαστε ότι παραμένουν κάποια λεπτά ζητήματα να επιλύσουμε δεν έχει νόημα. Γιατί δυστυχώ όλα τα παραπέμπουμε στις τεχνικές συνεδριάσεις και δεν καταφέρουμε να βγάλουμε άκρη. Για τους σκοπούς να σας πω ότι σκοπός μου ήταν να εισαγάγω ένα στόχο προκειμένου να υπάρχει ευθύνη. Να σας ευχαριστήσω για την κυρία Ρανς Γκαρσία. Ξέρω ότι δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Προσπαθείτε ως ομάδα να τα ρυθμίσετε αυτά καλά. Αλλά θεωρώ ότι όλο και πιο πολύ απέχουμε. αν ε, υπάρχουν κάποιες ε, περιοχές οι οποίες μόνιμα δεν θα καλλιεργούνται, για παράδειγμα. Κάποιοι πούνε ότι ναι, κάποιοι άλλοι ενδεχομένω να λένε ότι η αλλαγή των καλλιεργιών είναι κατηφετικό. Αυτό δεν ε, αλλάζει, δεν μπορεί να συνάδει ως τεχνική, αλλά αυτό δεν το παίρνουμε υπόψη, δεν συμφωνούμε, γιατί δεν θα συμφωνήσουμε ούτε σε 5 χρόνια, ούτε σε 10 χρόνια και σε άλλες επιφάνειες και καλλιεργίες. Δεν συμφωνούμε. Τι γίνεται, για παράδειγμα, για νέες ε, καλλιεργίες, για νέες ε, επιφάνειες καλλιεργίες. Ακόμα και για τέτοια θέματα δεν συμφωνούμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα απλά να πω στους συναδέλφους από την Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων ότι κοιτάξτε, έχουμε κάθε καλή διάθεση, αλλά απέχουν τόσο πολλοί οι απόψεις μας που δεν ξέρω κατά πόσον θα καταφέρουμε να βρούμε τελικά κάποιο συμβασμό, τον οποίο να προσυπογράφουν διάφορες πολιτικές ομάδες. Ο πρόεδρος. Ναι, αλλά όπου υπάρχει θέληση και όπου υπάρχει και σκληρή δουλειά, υπάρχει δυνατότητα και ελπίδα για να βρούμε ένα κοινό δρόμο. Αν ε, υπάρχει τρόπος να τον βρούμε. Ο κύριος Νίκολσον. Σα ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Α, συγγνώμη, σας ευχόμαστε και χρόνια πολλά. Είναι τα γενέθλιά σας. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε ότι όταν φτάνει κανείς αυτή την ηλικία προτιμά να τα ξεχνάει τα γενέθλιά του. Τι να κάνουμε, δεν θα αποφεύγει κανένας όσο πέραν τα χρόνια να ξεκινήσω λέγοντας ε, ότι η συγγετρία έχει πάρα πολύ σκληρή δουλειά να κάνει, πάρα πολύ δύσκολη σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες αυτές που ε, έλαβε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι είναι πραγματικά τιτάνιο το έργο το οποίο έχει κάνει ως τώρα. Και πιστεύω ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το θέμα λοιπόν η ΚΑΠ είναι ε, μια διαδικασία. Έχω παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία σε βάθο χρόνου. Θα πρέπει να την εξετάσουμε λοιπόν ως μια διαδικασία την όλη πολιτική. Μια διαδικασία που βελτιώνεται. Κάθε φορά που γίνεται η μεταρρύθμιση κάπου γίνεται και μια βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή ως ε, εισηγητέ και ως κοιόδες εισηγητέ. Αυτή είναι η πρόκληση λοιπόν που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πολύ χρόνο έχουμε δαπανίσει και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη του προσωπικού και τους βοηθούς που το κάνουν αυτό. Αυτό το οφείλουμε, είναι καθήκον μας και προς τους αγρότες αλλά και προς τους καταναλωτές γιατί αν δεν υπήρχαν αγρότες δεν θα υπήρχαν και τρόφιμα για τους καταναλωτές. Αυτή είναι λοιπόν η πρόκληση στην οποία θα πρέπει να τα εδώ στην Επιτροπή μας. Θα το και καιρό άλλωστε. Και αυτό πρέπει να το εξηγούμε συχνά σε άλλε επιτροπές και σε άλλου ανθρώπου. Ο σκοπό λοιπόν τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ είναι να διορθώσουν τα λάθη του παρελθόντο. Ένα από τα βασικά ζητήματα λοιπόν είναι το εξή. Συζητάμε μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ χωρί να ξέρουμε όμω πώ θα διαμορφωθεί τελικά ο προπολογισμό. Δεν έχει νόημα λοιπόν να πισωγυρίζουμε και να ακούμε διάφορα επιχειρήματα, γιατί μέχρι ότου ενημερωθούμε για τον προπολογισμό, που θα είναι μάλλον στο επόμενο κοινοβούλιο, δεν θα μπορέσουμε να ξέρουμε ακριβώ τι γίνεται. Να σα πω λοιπόν ότι μέχρι ότου διευκρινίσουμε τον προπολογισμό, δεν ξέρουμε τι έχουμε να δαπανίσουμε. Η γεωργία λοιπόν θα πρέπει να είναι σταθερή. Πρόκειται για αυτή είναι η βασική αρχή της ε, γεωργικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στρατηγικά σχέδια είναι πραγματικά το περιεχόμενο τη ε, μεταρρύθμιση. Θα πρέπει λοιπόν να τα διαμορφώσουμε με σωστό τρόπο για του γεωργού μα και θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε του γεωργού να παράγουν τελικά σωστά τρόφιμα για το λαό τη Ευρώπη. Αυτή είναι η βασική πρόκληση. Επίση, θα πρέπει να μπορούμε να δημιουργήσουμε τελικά μια πολιτική η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τι περιβαλλοντικέ ανάγκε τη Ευρώπη. Εγώ πάντα λέω ότι η Ευρώπη και η γεωργία δεν είναι θέμα του περιβαλλοντικού προβλήματος της Ευρώπης. Είναι το τμήμα της λύσης του προβλήματος και αυτό φαίνεται σε όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα να το γνωρίσουμε πιο πολύ αυτό. Μέχρι ότου το γνωρίσει πιο πολλοί κόσμος λοιπόν αυτό δεν θα βρούμε μία λύση. Δεν έχει νόημα να δακτυλοδεικτούμε ή μέντος δε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας η πολιτική αυτή και αυτό είναι που μας διακρίνει στην Ευρώπη. Αυτό και θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Όπως είπε και ο Επιτρόπος Όγκαν σε διάφορες περιστάσεις, η ανάγκη για την απλοποίηση υπάρχει. Άκουσα διάφορα επιχειρήματα για την απλοποίηση εδώ στην Επιτροπή σε διάφορες περιστάσεις και πιστεύω ειλικρινά ότι με τα μεταρρύθμιση αυτή Και ειλικρινά, ακούγοντα μερικού ανθρώπου να μιλάνε, έχω την εντύπωση ότι έτσι όπω τα λένε μερικοί, αν ακολουθούσαμε την άποψή του, θα είχαμε πιο πολύ γραφειοκρατία τελικά, όχι λιγότερη. Και θα χανόμασταν σε κικαιώνε. Καταλαβαίνω, Πρόεδρε, ότι θέλω να πάρω το λόγο κι άλλοι. Αναγνωρίζοντας ε, τους στόχους και των άλλων ομάδων, θα πρέπει να διακρίνουμε και ποια είναι η διάθεση που επικρατεί και να πετύχουμε και καλά αποτελέσματα. Να σας πω ότι η μεταρρύθμιση δεν θα ολοκληρωθεί στο κοινοβουλίο αυτό, αλλά αυτό που θα πετύχουμε θα πρέπει να περάσει στι διαπραγματεύσει. Θα πρέπει να μπουν λοιπόν και στοιχεία τα οποία να μπορούμε να τα θυσιάσουμε. Και ελπίζω η συγκήτρια να παραμείνει και στο επόμενο κοινοβούλιο για να μπορέσει να το προχωρήσει το θέμα αυτό, γιατί έχει πραγματικά πολλή εμπειρία τα πιο πολλά στοιχεία τα οποία μπορεί να τα διαπραγματευτεί στην ανάλυση. Γιατί τελικά αυτό θα γίνει για να αποτύχουμε το τελικό πακέτο. Για τους γεωργούς. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Οι μεταρρυθμίσεις πάντα αποτελούν ενός είδους προσαρμογή Γι' αυτό λοιπόν και έχουν τέτοιο μεταεξελικτικό χαρακτήρα. Σε ό,τι τον προπολογισμό, δεν θα είναι πιο χαμηλό από αυτόν που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Χάιτομα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να συνεχίσω ε, αυτά που πήγε να πει ο κύριος ε, Νίκολσον. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η πορεία και μετά τις ε, εκλογές ε, με την επανεκλογή γιατί πρόκειται για τεράστια προσπάθεια τους ώστε να κλείσουμε το θέμα στην πρώτη ανάγνωση. Ο εχθρό εδώ είναι το ρολόι, ο χρόνος, κρίμα. Γιατί έχουμε πάρα πολλές δυσκολίε, πάρα πολλές αντιρρήσεις, αλλά τελικά οι διαφορές μας δεν είναι τόσο μεγάλες θέλουμε να πετύχουμε στο μέτωπο του ανταγωνισμού, στο μέτωπο του περιβάλλοντος, στο, να, έχουμε κάποιο είδους ε, κάπου που να είναι απλή, μην είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και α, άλλα σκηνού φυσικά στη Βλανδία από ό,τι στην Νότια Πορτογαλία. Έχουμε την πρόταση της Επιτροπής, και ίσως το πρασίνισμα σήμερα δεν έχει πετύχει, αλλά ίσως θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τα αποτελέσματα και όχι στο να εξετάζουμε τα μέτρα και να ληφθούν μέτρα που να ισχύουν για όλους. Να πιάνουν τόπο προσπάθεια στον Γιώργο, να υπάρχουν αποτελέσματα. Μπορούν όλες οι πολιτικές ομάδες να δουν την πρόταση ίσως με άλλο δρομολόγιο κάθε ομάδα, γιατί μερικές ομάδες θέλουν να υπάρχει περισσότερη ρεσιμότητα, αλλά επίσης δεν θα πρέπει να πιεντρωνόμαστε πάρα πολύ στα μέτρα, να έχουμε περισσότερη ευελιξία. Ας κοιτάξουμε καλύτερα τα αποτελέσματα, τους στόχους σε σχέση με αυτήν την αναβαθμισμένη ε, Εγώ, ας πούμε, θα υπάρχει αυτού του είδους το οικολογικό πρόγραμμα, άλλοι θέλουν δεύτερο πυλώνα. Εντάξει, σου πω την αλήθεια, δεν με νοιάζει πώς θα το πετύχουμε, αλλά βλέπω ότι έχει μια θετική τάση. Είναι μια ευκαιρία το ότι όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, να κάνουμε την πιο αποτελεσματική, πιο απλή, πιο αποτελεσματική και να πετύχουμε και για το πρασίνισμα και για την ανταγωνιστικότητα. Άρα, ελπίζω τι αμέσω σε επόμενε μέρε και εβδομάδε να τα πετύχουμε και να καταλήξουμε σε μια αρχιτεκτονική που θα αρέσει σε όλου. Χόσλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, αλλά νομίζω ότι πήγαμε σε άλλη εκδήλωση. Δεν είχα την εντύπωση ότι προχωρήσαμε καλά. Από όλε αυτέ τι ε, τροπολογίε που έχουμε να επεξεργαστούμε, είναι τόσο πολλέ και διαφορετικέ οι απόψει που επικρατούν, που δεν ξέρω πώ θα καταφέρουμε να τι επεξεργαστούμε. Είπατε ότι. Μάλλον έχουμε μία άποψη κι εμεί, έχει και μία άποψη η συγγήτρια. Τώρα, κατά πόσο αυτή είναι η άποψη όμω του ΕΛΚ, δεν το ξέρουμε. Μπορούμε να το λέμε. Αλλά ψηφίσαμε και την έκθεση Ντόρφμαν, που κινήθηκε προ διαφορετική εντελώ κατεύθυνση. Μου προκαλεί λοιπόν εντύπωση το γεγονό ότι μα λέτε ότι αυτή είναι η άποψή μα και μα υποστηρίζουν και δύο άλλε πολιτικέ ομάδε. Εγώ έχω την εντύπωση στι διαπραγματεύσει ότι και από πλευρά μεθοδολογία υπάρχουν αμφιβολίε. Πάμε σε όλε αυτέ τι τεχνικέ συνεδριάσει. Ωραία, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε 12 τεχνικέ συναντήσει που παίρνουν από μισή μέρα και δύο συνεδριάσει σκιωδών που παίρνουν δύο ώρε. Και Υποτίθεται ότι όλα τα πολιτικά ζητήματα θα τα έχουμε επιλύσει μέσα σε δύο ώρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τόσο πάρα τα πολιτικά ζητήματα που θα αποκλείεται. Αυτή είναι η διαφορά με αυτά που είπε η κυρία Μούλερ. Ότι κοιτάμε τι ε, παραγράφου μία προ μία, αλλά δεν κοιτάμε κατά πόσον όλο το σύστημα τελικά είναι σωστό. Για παράδειγμα, η έκθεση Ντόρτμαν δεν είναι αυτό που θέλουμε ω κοινοβούλιο δεν μπορούμε να κοιτάμε παράγραφο όπως παράγραφο το κείμενο και να λέμε «Ε, εντάξει, κάπου τα βρήκαμε». Στην ψηφοφορία τελικά θα γίνει χαμός, γιατί δεν ταιριάζουν όλα αυτά τελικά μεταξύ τους. Και μόνο και μόνο το θέμα των προδιαγραφών. Πόσο δεσμευτικές είναι, πόσα χρήματα μπαίνουν και πηγαίνουν στο θέμα αυτό. Ποια είναι η χρηματοδότηση λοιπόν. Αν δεν ξέρουμε ποια είναι η χρηματοδότηση, πώ θα τα διευκρινίσουμε όλα αυτά. Ο δεσμευτικό χαρακτήρα του δεύτερου πυλώνα. Δεν ξέρουμε αν ο πρώην δεύτερο πυλώνα τελικά έχει χρήματα, πόσο χρήματα έχει. Όλα αυτά λοιπόν δεν μα επιτρέπουν να μπούμε σε επίπεδο λεπτομέρεια ή, εν πάση περιπτώσει, όχι στο επίπεδο λεπτομέρεια που θέλει η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή, αυτή, η, συγγνώμη, η συγγνωμη η στην παρούσα φάση. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι θα προκληθεί μεγάλη σύγχυση. Αναφέρθηκε αυτό και εγώ. Ακόμα και ορισμός των, ε, του βοσκοτροπιού δεν ε, μας βρίσκει σύμφωνος. Χάος θα προκληθεί. Γι' αυτό λοιπόν αναρωτιέμαι πώς τελικά θα, θα συζητήσουμε όλα αυτά, πώς θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Γιατί θεωρώ ότι το χειρότερο δυνατό σενάριο θα ήταν να υποβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια εντελώ ανώριμη πρόταση και να κληθούμε να συζητήσουμε το Συμβούλιο, το οποίο θα τα απορρίψει όλα αυτά παρά αυτά. Νομίζω ότι η ενίσχυση του Κοινοβουλίου και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το πιο βασικό στοιχείο. Και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε την εργασία μας όπως ε, Ω τώρα δεν θα πετύχουμε μια ισχυρή τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε μέχρι το τέλο τη αιτία. Ήδη έχουμε καταφέρει αρκετά και τώρα πάντω θα πρέπει οι προσπάθειέ μα να αποδώσουν καρπού. διότι θα πρέπει να λογοδοτήσουμε στου ψηφοφόρους. Θα μας ρωτήσουν τι καταφέρατε, τι κάνατε. Όλοι για την ε, ΚΑΠ κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ό,τι καλύτερο. Και έχουμε συζητήσει και το θέμα της βελτίωσης της ΚΑΠ. Οπότε προκειμένου θα πρέπει να είμαστε αυστηροί γιατί αυτό θα βοηθήσει. Αλλά βέβαια να μην καταλήξουμε σε κατάσταση χαοτική. Κύριε Φλάναγκαν, ευχαριστώ. Σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Γκαρθία, τα άκουσα. Αυτά που είπατε στα αγγλικά και η μητρική μου γλώσσα, αλλά δεν τα κατάλαβα καλά. Τι είπατε, ότι θα πρέπει να βιαστούμε και ο κόσμος θα καταλαβεί τότε γιατί δεν αρχίζαμε πιο νωρίς για να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος. Σπέβδε βραδέως λέμε και άρα θα πρέπει για κάτι τόσο σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί. Πάντως για μένα και για τους εφόρους μου το πιο σημαντικό είναι και νόμιζα ότι και για το ΕΛΚ και για το δικό μου κόμμα είναι το πιο σημαντικό να υπάρξει το 2026 100% σύγκληση. Σύμφωνο. Δεν είναι εδώ να συνεχίσουμε να πληρώνουμε για, κάτι το οποίο έγινε πριν από 20 χρόνια. Αν έχουμε 75% σύγκληση το 26, τότε δεν κάνουμε τίποτα προτιμώ να μου πείτε την αλήθεια. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Λέμε για τη βιωσιμότητα και την αναδιανομή των πόρων μετά το κάπινγκ. Θα δούμε τι λένε οι οικονομολόγοι που είναι ειδικοί στη Γεωργία, όπως ο Μάθιος. Θα δούμε πώς το κρίς θα γίνει πιο ανθρώπινο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα προσφυγών. Το έχω μελετήσει. Αυτό, το, αυτός ο λόγος είναι ο βασικός λόγος που ο κόσμος έχει γίνει προσκεπτικιστής. Το Ντόνεγκαλ έτσι λένε, υπάρχει οργή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πάρα πολύ αυτοί που ασχολούνται με το περιβάλλον. Και όταν απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρωτήσουν αν τα πράγματα πάνε καλά, ε, αν έχει γίνει σωστή ρύθμιση για τη χώρα τους, τότε τους θέλουν από τον Άννα στον Καϊάφα. Υπάρχει απάντηση. Αν είναι να πάμε για τα στρατηγικά προγράμματα, να υπάρχει κάποιο δεύτερο μορφό δικαιοδοσία, κάτι σαν προσφυγή για να πάει ο κάθε Γεωργό και να αισθάνεται δικαιοσύνη. Τα είδαμε στην, ε, στην πρόταση τη σχετική που έγινε στον έλεγχο των προπολογισμών σήμερα το πρωί και πέρασε. Άρα αφογκραστείτε αυτού του ανθρώπου. Δεν είναι δυνατόν εδώ να ζούμε σε βένινο πύργο. Να ακούμε τι λέει ο κόσμο. Αυτό είναι ο βασικός λόγος που έχουμε περικοπεί στην ΚΑΠ. Γιατί στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού λένε ότι τα πράγματα μπορούν να συνεχιστούν έτσι. Δεν πάνε τα λεφτά εκεί που πρέπει. Εμείς όμως τους δίνουμε ε, λαβή για να κάνουν την περικοπή. Δεν πρέπει να στριμώχνουμε, να τιμωρούμε τους Γιώργους δεν κάνουν αυτό που του ζητήσαμε. Τώρα για του νέου γεωργούς θα πρέπει να μπορούν να αναλάβουν την εκμετάλλευση όταν, ε, όταν μπορούν. Στο 6.1G λέει ότι αυτό είναι συγκεκριμένο στόχο. και από την εμπειρία μου από την προηγούμενη μεταρρύθμιση αυτή η διατύπωση αυτό το οποίο λέμε πρόσφατα στημένη, πρόσφατα συγκροτημένη, είναι κακό για το στόχο. Έχω και άλλη τροπολογία που έχω υποβάλει σε σχέση με την αλλαγή από εκεί που λέει ε, δεξιότητες ε, υπάρχουσες σε δεξιότητες ε, αποκτώμενες. Και έτσι να πάμε για επίτευξη του στόχου για το περιβάλλον. Έχουμε κάποιο σχετικό πρόγραμμα στην Ιρλανδία αλλά και στην Ισπανία. υπάρχει βαθμολόγηση που έχει πετύχει ο καθένας και αμείβεται αναλόγως ο πρόεδρος. Κυρίε και κύριοι, και τώρα έχει ο καθένας δύο λεπτά στη διάθεσή του, διότι αναλώσαμε το χρόνο των σκιωδών Κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους κοιόδες εισηγητές. Δεν θα ήταν εύκολο, το ξέραμε. Και βλέπω ότι είναι περίπλοκο. Ναι. Καταλαβαίνω ότι παραμένει περίπλοκο το θέμα. Δεν είναι εύκολο, κυρίως γιατί δεν πρόκειται απλώς για μια νέα μεταρρύθμιση, αλλά για μια μεγάλη αλλαγή. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, η οποία γίνεται, αλλά είναι περίπλοκο. Η συζήτηση δεν μου άρεσε που λέγαμε αυτή η πολιτική ομάδα θέλει αυτό, η άλλη πολιτική ομάδα θέλει το άλλο. Η δικιά μου η πολιτική ομάδα δεν έχει την ίδια άποψη για πολλά. Για άλλα συμφωνεί, για άλλα δεν συμφωνεί. Δεν ε, λειτουργούμε ως μπλοκ και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει με όλους και με το ΕΛΚ. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Συνεπώς, Έχουμε κάποιες γραμμές βέβαια κατά προτεραιότητα που στηρίζουν οι συγητές μας, ναι. Αλλά δεν μου αρέσει να καθόμαστε και να συζητάμε βάζοντας αντιπαράθεση τη μία ομάδα με την άλλη. Σε ποια θέματα θέλω να σταθώ. Το συνδυτοποιούμε ότι πολύ σύντομα θα ψηφίσουμε. Και μετά να κάνουμε γασπάτσο, μια κρύα σούπα έτσι σπανική γασπάτσο, να το απολαύσουμε. Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε όλοι ό,τι περνάει από το χέρι μας, παρόλο που είναι περίπλοκο το θέμα. Λοιπόν, κύριε Ράντς και στους κοιόδης συζητητές θέλω να τα πω. Συγκεκριμένα, για το κάπινγκ, το ανώτατο όριο. Για τη δικιά μου πολιτική ομάδα είναι σημαντική κόκκινη γραμμή. Είναι υποχρεωτικό. Ξέρω ότι για σας όχι, για μας ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρω ότι κάνουμε υποχωρήσεις. Γιατί δικαιολογούμε να υπάρχει μια εκμετάλλευση που να παίρνει 600.000 ενισχύσεις, μόνο ενίσχυση και να δημιουργεί το χρόνο 23 θέση απασχόληση, το λέω γιατί έχω τέτοια περίπτωση, την ξέρω. Δικαιολογείται αυτό? Όχι για μένα. 600.000 ευρώ. Γι' αυτό θέλω κάπινγκ ανώτατο όριο. Γιατί θέλω να υπάρχει ένα όριο στις ενισχύσεις της εκμεταλλεύσεις. Με 23 υπαλλήλου και 600.000 ευρώ, ε, πώς σας φαίνεται. Αυτό το μοντέλο θέλουμε. Όχι. Πέρα από το μοντέλο όμως, τα λέω, γιατί τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν με τη σημερινή ΚΑΠ και στη δική μου περιφέρεια και αλλού. Οπότε, να, να μου εξηγήσουν αυτοί που δεν θέλουν το κάπινγκ, γιατί. Εγώ θέλω καλύτερη αναδιανομή οι συνδεδεμένες πληρωμές. Πιστεύω ότι είναι κάτι σημαντικό, αλλά προσοχή και εδώ. Όχι ο καθένας για το χωριό του, έτσι. Προσοχή. Αυτά τα πράγματα εγώ τα βλέπω να συμβαίνουν. Μην μπερδεύουμε και ανακατεύουμε λάδι, κρασί και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, συνδεδεμένες πληρωμές, αλλά εκλογικευμένες, είτε πρόκειται για το κρασί, το μέλι, δεν ξέρω πρέπει να βάλω και το λάδι εδώ. Έπειτα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, και τελειώνω, συγγνώμη μακρηγορώ, πρέπει να προσθέσουμε και άλλη ενισχυμένη αιρεσιμότητα προϋπόθεση δηλαδή. Δεν πρέπει να είναι σε χειρότερη θέση μία εκτενοτροφική εκμετάλλευση εξαιτία των συνδεδεμένων ε, ενισχύσεων. Ξέρω ότι κυρία Ρένς και εσείς και οι σκιώδες εισηγητές ε, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι Δεν λέω ότι εγώ θα τα κατάφερνα καλύτερα, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Και αν σε πέντε εβδομάδε τα καταφέρουμε, τόσο το καλύτερο. Γιατί πρέπει να ψηφίσουμε σε πέντε εβδομάδε, έτσι. Πρόεδρο, πέντε λεπτά ήταν. Πώ θα είμαι αυστηρό τώρα με του υπόλοιπου. Δεν είναι δυνατόν να αναπτύσσετε τις θεωρίες σας για δύο λεπτά και μετά κάνετε ερωτήσεις. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Σερδός. Πρώτα απ' όλα να πω ότι υπάρχει μια λύση πάνω στην οποία έχω δουλέψει εγώ και αυτό είναι η μερική μείωση σε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πουλερικά, αυγά. Επίσης, περιλαμβάνοντας αυτούς τους κανόνες τώρα και αυτό νομίζω ότι είναι θετικό. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καθορίσουν δίκτες επιδόσεων. Και το ίδιο και για την ερεσιμότητα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να φροντίσουν για τους κανόνες της χώρες μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να έχει δικαιώματα εξουδιωτικών ε, πράξεων. Έπειτα, η στήριξη Έχουμε πολύ ευαίσθητους τομείς όπως είναι το πρόβιο, το έγιο κρέας. Πρέπει αυτούς τους τομείς να τους ενισχύουμε και θα ήθελα αυτό να το δω στο κείμενο. Και τρίτον, η στήριξη για τους νέους αγρότες. Η συγγήτρια πρότεινε 3% αρχικά. Εγώ θέλω να το στηρίξω. Γιατί δεν έχουμε την νέα παραγωγών πρέπει να τους στηρίξουμε. Θα πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους μας αυτό. Το 2% δεν φτάνει για τις άμεσες ενισχύσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι 3%. Το ελάχιστο αντί για το 2%. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Κατάινεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές έχετε εργαστεί με πολύ σφιχτές προθεσμίες, το ξέρω. Ωραία, και τώρα θα μετρήσω το χρόνο μου για να μην μακρηγορήσω. Λοιπόν, θέλω να τονίσω κάποια πράγματα ε, που ζητάω από τους κοιόδους εισηγητές να λάβουν υπόψη τους όταν να καταρτήσουν συμβαστικές τροπολογίες. Τα οικολογικά σχέδια και ρεσιμότητα είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε συνολικά δεν πρέπει να είναι πολύ αυστηρά ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γιατί θα φέρουν παραπάνω προβλήματα στους παραγωγούς. Γιατί τότε η κοινή γεωργική πολιτική δεν θα εξυπηρετεί το σκοπό της. Αν καταλήξουμε σε πολύ αυστηρά μέτρα για τα οικολογικά προγράμματα, δεν τα καταφέρουμε. Πρέπει να δώσουμε ευελιξία στις χώρες μέλη για να υλοποιήσουν τέτοια μέτρα, όπως και για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Οι χώρες μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα μέτρα όσο καλύτερα ε, για την δική τους την κατάσταση, σύμφωνα με τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Θέλω να σας δώσω ένα Παράδειγμα για το GAEC2. Στις βόρειες χώρες υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσει από τις άλλες. Και αυτό γιατί το μεγαλύτερο τμήμα των ορόσημων γεών μας είναι με τύρφη. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ευελιξία και να μην είμαστε πολύ αυστηροί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, The most Συμφωνώ και με την εκτίμηση ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η επόμενη θητεία τελικά θα κληθεί να αποφασίσει για το θέμα αυτό. Αναφέρθηκε το θέμα του προπολογισμού. Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα σενάριο που το ΚΑΠ, το προπολογισμό που θα μειωθεί κατά 50% σε μια συνολική αύξηση του προπολογισμού. Εγώ ελπίζω ότι η ίδια μου η κυβέρνηση δεν θα προσυπογράψει το σενάριο αυτό. Και οι άλλες, ε, και οι άλλοι θα καταψηφίσουν μια τέτοια γέλια άμα, πρόταση. Μέχρι ότου λοιπόν ε, οριστεί ο προπολογισμό, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να, ορίσουμε τη νέα πολιτική. Στο πλαίσιο του περιορισμένου χρόνου που έχω στην διάθεσή μου και σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, πιστεύω ότι ναι, θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία πόρων και μια αναδιανομή. Είναι πραγματικά... Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα σύστημα που θα καταπνίξει ένα σύστημα το οποίο υποστηρίζει τους αγρότες που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Είναι πραγματικά ηθικά παράδεκτο κάτι τέτοιο. Και είναι ένα από του λόγου για του οποίου είναι δύσκολο να εξηγήσουμε τελικά στου καταναλωτέ σε όλη την Ευρώπη γιατί η κοινή γεωργική πολιτική είναι τόσο σημαντική. Χρειαζόμαστε την κοινή γεωργική πολιτική να λειτουργεί. Αν θέλουμε να έχουν κάποιο μέλλον αυτές οι κοινότητες. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο είναι διαφανές και το οποίο δεν πιστεύεται ο κόσμος και πάνω απ' όλα να είναι ένα σύστημα το οποίο τελικά θα λειτουργεί για αυτούς που παράγουν τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουν οι καταναλωτές. Κορυφαία ποιότητα σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει αναδιανομή των πληρωμών για, τον, για τους ανθρώπους αυτούς που υποστηρίζουν τελικά το σύστημα παράγοντα το τρόφιμα που καταναλώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στουσάντος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Να ευχαριστήσω την κυρία Αγγιλέρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, μιλάει για πιο πολύ ευελιξία για τα κρατημέλη σε ό,τι αφορά διάφορες παρεμβάσεις που πιστεύουν ότι ταιριάζουν πιο πολύ στις ανάγκες μας. Αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που θα αντικατασταθούν από εθνικές προδιαγραφές και από τοπικές προδιαγραφές δεν είναι προφανώς κατευθυντικό αυτό, γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Είναι διαφορετικέ οι βασικέ δραστηριότητε, οι αγροτικέ δραστηριότητε και δεν συγκρίνονται με αυτέ άλλων ε, ήπειρων. Θα πρέπει να γνωρίσουμε λοιπόν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφορών περιοχών σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό θα μπορέσουν ε, οι περιφέρειες να θέσουν ε, τις ε, διαγραφές που χρειάζονται για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ο κ. Ροπέ. Να ευχαριστήσω και εγώ και να συγχαρώ την συγκέντρια. Ήταν πραγματικά Ηράκλειο το έργο. Και Μάλιστα και εγώ ασχολούμαι με το θέμα αυτό στα πλαίσια της Επιτροπής Περιφερειακής ανάπτυξη. Κατανοώ λοιπόν ποιε είναι οι προκλήσει. Φυσικά δεν θα πρέπει να βιαστούμε, θα πρέπει να δώσουμε χρόνο στην ε, πρόταση αυτή. Είναι πολύ σημαντική για το μέλλον μας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε ασάφεια, οποιαδήποτε ασυμβατότητα στο έγγραφο αυτό. Κατανοούμε λοιπόν ότι το Συμβούλιο δεν ε, θα το εξετάσει το έγγραφο αυτό πριν από το φθινόπωρο. Έχουμε λοιπόν χρόνο να προσπαθήσουμε να συγκλίνουμε τις απόψεις μας. Για να πετύχουμε πραγματικά από τα αποτελέσματα. Ένα θέμα λοιπόν είναι και η εξωτερική σύγκληση. Η ΚΑΠ αποτελεί μία και μόνο πολιτική για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ίδιες προδιαγραφές για όλους. Η υποστήριξη όμως διαφέρει δεν είναι λοιπόν εύκολο να συναγωνίζονται διάφοροι αγρότες για τέτοια θέματα στην ενιαία αγορά. Είναι αδύνατον. Και νομίζω ότι έχουμε έρθει σε ένα σημείο που πρέπει να ολοκληρώσουμε πραγματικά τα θέματα αυτά. Σήμερα λοιπόν. Μιλάμε για ένα τρέχον μέσο όρο το οποίο θα έπρεπε να λάβουν όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να ορίσουμε λοιπόν τους κανόνες και τις ημερομηνίε με σαφήνεια. Πότε θα πετύχουμε την πλήρη σύγκληση προκειμένου όλοι να συναγωνίζονται επίσης ώρες. Όχι μόνο οι αγρότες αλλά και τα κράτη-μέλη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίφαση η οποία θα παραμείνει και στο μέλλον. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Έχουμε διάφορες λοιπόν προτάσεις. Ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποια κοινά σημεία, τα οποία να είναι αποδεκτά για όλους. Ευχαριστώ κυρία Σολάνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. συγχαρώ την εισηγητρία και του συνεισηγητέ. Ξέρω ότι έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και ότι είναι πολύ διαφορετικέ και αποκλίνουσε οι απόψει. Ακόμα και μέσα στην ίδια πολιτική ομάδα. Θα ήθελα να υπάρχει μια ισορροπία και να λάβουμε υπόψη ναι, οι ιδιαιτερότητε τι ιδιαιτερότητε τη γεωργία σε κάθε χώρα. Να ξεκινήσω από ένα θέμα όπου η άποψή μου διαφέρει από την ε, άποψη της ομάδας μου σε ό,τι αφορά το κάπινγκ, τα ανώτατα όρια. Δεδομένων λοιπόν των συγκεκριμένων ε, χαρακτηριστικών της γεωργίας σε κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μου χώρα, η, Ρωμανία... δεν ε, θέλουμε να υπάρχει ουσιαστικά ανώτατο όριο. Δεν θέλουμε να υπάρχει κάπινγκ. Αν στη συνέχεια επιβληθεί κάποιο κάπινγκ, θα πρέπει να είναι εθελούσιος ό,τι αφορά τις ε, πληρωμές διανομής. Συμφωνώ ότι οι μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης. Όταν μιλάμε όμως για τα ανώτατα όρια, ιδιαίτερα για το επίπεδο του κάπινγκ που μιλάμε σήμερα, μιλάμε ουσιαστικά για μεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί η γεωργία η οποία οδηγεί στην παραγωγή τροφίμων ουσιαστικά βασίζεται στις μεγάλες και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε τρόπους να υποστηρίξουμε και τους μικρούς γεωργούς. Αλλά δεν θα πρέπει στη διαδικασία αυτή να ξεχνάμε τι γίνεται και με τις μεσαίες και μεγάλες ε, επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους νεαρούς γεωργούς και στο σημείο αυτό θα κλείσω. Συμφωνώ ότι 3% για άμεσες πληρωμές είναι ένα σωστό ποσοστό. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους νεαρούς γεωργούς, τους χρειαζόμαστε στην Ήπεθρο, ιδάλλως έχουμε το θέμα της αστιφιλίας, το οποίο κανείς δεν το θέλει για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σχράιερ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ κατέθεσα τροπολογίες, 70. για τους ε, γεωργούς και για τις ε, περιοχές. Σε ό,τι αφορά τις άμεσες επιδοτήσεις ε, θα πρέπει να έχουμε ή συνταμιβή για τις υπηρεσίες που μας δίνουν οι γεωργοί. Οι κρατικοί κανόνες και η γραφειοκρατία όμως εμποδίζουν αυτή την πρόταση. Η προϋπόθεση είναι λοιπόν να υπάρχουν, να αφαιρεθούν οι περιορισμοί. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να δώσουμε 30% του πρωτοπυλώνα για τους γεωργούς, παρά το γεγονός ότι τα βοσκοτόπια συμπεριλαμβάνονται στον Natura 2000, αν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Δεν είναι δυνατόν όμω να το επιτρέψουμε αυτό. Μιλάμε για νέα συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακούει την Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων και τι συζητήσει μα, ή μήπως συνεχίζει και κάνει του κεφαλιό τη. Ευτυχώς κατάθεσαν όλοι οι συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά την ε, απαγόρευση ε, δοκιμώνα, ε, θεωρώ ότι αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα χωρίς να προαγάγει τίποτα στις τροπολογίες 51-59. Να κοιτάω ακριβώς το θέμα της Natura 2000. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση. Ελπίζω ω ε, βουλευτέ να μπορέσουμε να στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διαφορά του νεαρού γεωργού. Προτείνω λοιπόν 33% τουλάχιστον από τον ε, πρώτο πυλώνα για τους νεαρούς ε, γεωργούς. Και σε σχέση με αυτά που είπε και ο κύριος Φαντεκάντελαρε. Ο κύριος Ντόρφμαν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω κάπως την εντύπωση στη συζήτηση αυτή ότι κάνουμε και υποκρινόμαστε ότι όλα είναι στραβά και ανάποδα. Μα δεν είναι ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε σήμερα μία ε, γεωργική πολιτική η οποία λειτουργεί. Κοιτάμε τώρα πού μπορούν να γίνουν βελτιώσει. Πού έχουν γίνει αλλαγέ ε, με την πάροδο του χρόνου που δεν είναι πλέον αποδεκτέ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επηρεαζόμαστε πολύ από αυτούς που εκμεταλλεύονται το σύστημα στην παρούσα φάση. Να μην χάσουμε και τον απόλυτερο στόχο. Γιατί ο απότερος στόχος είναι να διατηρηθούν τελικά οι οικογένειες γεωργών στην Ευρώπη και να παραμείνει ζωντανή η ύπεθρος. Αυτό λοιπόν πατυχαίνουμε με τον πρώτο πυλώνα. Στον πρώτο πυλώνα, με την πάροδο του χρόνου, ε, έγιναν διάφορες εξελίξεις οι οποίες πλέον δεν στέκουν. Έχουμε δικαιούχου που δεν είναι γεωργοί, που δεν έχουν ουσιαστικά να κάνουν τίποτα πλέον με τη γεωργία. Παίρνουν όμως κάθε χρόνο τα χρήματα. Με την ε, κοινή ερωτική πολιτική κάνουμε ε, επενδύσεις και για επενδύσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι βλέπουμε. Βλέπουμε επενδύσεις που σε διάφορες περιπτώσεις δεν έχουν να κάνουν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι είναι λοιπόν καθήκον της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής ε, να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις ε, Ρώσων ή Αμερικανών. Αυτό το κάνουμε σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Βλέποντας λοιπόν ποια σφάλματα υπάρχουν, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι χρειαζόμαστε κάποιο κάπινγκ, χρειαζόμαστε νέο μοντέλο στον πρώτο πυλώνα, χρειάζεται μια καινούργια σύγκληση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τις πληρωμές που γίνονται σήμερα σε μη ενεργούς γεωργούς. Όταν λοιπόν αυτά καταφέρουμε να τα κάνουμε με έναν σωστό τρόπο, θα καταφέρουμε να βρούμε και μια καλή λύση για τη γεωργική πολιτική την επόμενη δεκαετία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Μας εξηγείτε ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι δοκιμασμένες λύσεις της ισχύουσας ΚΑΠ. Ναι, ναι. Βάιτς. Όπως βλέπουμε και στο ΕΛΚ υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Κάποιε ερωτήσει να κάνω στην εισηγήτρια. Τι εννοείται ακριβώ με τον πραγματικό αγρότη. Για παράδειγμα, κάποιο ο οποίο βγάζει λεφτά κατά 70% ε, από τον τουρισμό, αλλά παρόλα αυτά κρατάει ε, την αγροτική του εκμετάλλευση, θεωρείται πραγματικό γεωργό. Τι, είναι οι προτάσει για να αποτρέψουμε τη στρέβλωση τη αγορά και σε ό,τι αφορά την, την Ουγγαρία, την Τσεχία, την Αυστρία, πώς αποτρέπεται τη στρέβλωση της αγοράς και πώς εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν συγκρίσιμα κριτήρια στον ίδιο χώρο αν αποφασίζονται όλα αυτά σε εθνικό επίπεδο. Γιατί μιλάμε για κάπινγκ 150.000 ήταν 70-60.000 και θέλετε να κάνουμε μόνο κάποια διάκριση. Μα αυτό δεν είναι κάπινγκ. Σα παρακαλώ, μην υποκρινόμαστε και να μην ε, εξαπατάμε και αυτού που μα ακούν. Δεν πρόκειται πλέον για κάπινγκ και κυρίω ε, αν λάβουμε υπόψη και του ε, μισθού. Δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Για 90% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων δεν χρειάζονται καν 150.000. Είναι πολύ πιο χαμηλά. Θα πρέπει αυτού να υποστηρίξουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε. Δεν είπα τα πρώτα 120 εκτάρια. Αυτό τι θα γίνει, θα αφαιρεθεί από την έκθεση. Και το Jim Nicholson να πω το εξή. Καταρχά, Jim, ναι, η γεωργία είναι κατά τμήμα μόνο ε, τμήμα τη λύση. Εν μέρη μόνο τμήμα τη λύση. Η δική μου, α πούμε, εκμετάλλευση είναι μέρο τη λύση. Δεν είναι όμω όλε τι εκμεταλλεύσει μέρο τη λύση. Κάποιε επιχειρήσει είναι μέρο του προβλήματο. και να το αναγνωρίσουμε αυτό. Θυμάμαι την εξαιρετική δουλειά που κάναμε, αλλά η υπουργό Κέρστιγκερ χθε ήταν εδώ και μα έλεγε ότι θα διατηρήσει τον γεωργικό προπολογισμό. Αν λοιπόν αυτό περάσει θα αποτελέσει μια αρνητική επίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω πριν λήξει η θητεία θα αποφασίσουμε. Δεν φαίνεται κάτι εύκολο, αλλά ας προσπαθήσουμε. Δεύτερον, συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ το 15% περικοπή για τις ανάγκες της ε, υπαίθρου. Θα είναι λάθος. Θέλω να υπάρχει περισσότερη ευελιξία και επικουρικότητα απλούστερο το σύστημα και λιγότερη έλεγχη για τους γεωργούς. Βεβαίως είμαι υπέρ του μοντέλου της ε, οικογενειακής γεωργίας. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ο ορισμός του κάπινγκ. Σίγουρα και οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις είναι καλύτερες για το περιβάλλον να μην τις υποστηρίζουμε μόνο με τα λόγια, αλλά και μέσω του κανονισμού. Τώρα, για τους νέους γεωργούς που ξεκινάνε και αναλαμβάνουν κάποια εκμετάλλευση, το θέμα είναι αυτοί που μεταβιβάζουν την ε, ε, επιχείρηση, την εκμετάλλευση. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όμως ότι πολλοί αποκτούν μια εκμετάλλευση όταν είναι 55 ε, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Επίση, έχουμε μελετήσει για το πρόβλημα του πώ θα χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή επανάσταση στην Ήπεθρο για να υπάρχει κάποιο είδους ε, υποδομή, κάποιο είδους ανάπτυξη δεξιοτήτων, να υπάρχει περισσότερη κινητικότητα στην Ήπεθρο Ε, να, έχουμε μια προσέγγιση συνεταιριστικής ε, οικονομίας. Ε, χρειάζεται τέτοιες λύσεις ύπεδος για να επιβιώσει. Σας ευχαριστώ, κύριε Νταντέν. Μπράβο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Ράς. Μπράβο που μας άκουσε επί τρεις μήνες. Δούλεψε σκληρά για να καταλήξει σε αυτόν τον συνδεσμό. Συχνά μας κατηγορούν οι Γεωργοί ότι αλλάζουμε συνέχεια τη νομοθεσία. Έχουμε αυτόν τον ζώντιο κανονισμό και όντως έχουμε λάβει κάποιες ε, αποφάσεις για το βιβλιοκομικό τομέα, για τις συνδεόμενες ενισχύσεις και άλλα. Ναι, αλλά όλα αυτά τα μέτρα τώρα άρχισαν να εφαρμοζούνται. Και εμείς ξεκινάμε τώρα νέα τροποποίηση. Ε, προσοχή, μην πέσουμε σε καμία παγίδα. Ας ε, μάθουμε από αυτά που έχουμε ήδη θεσπίσει. Και βέβαια να απολαύσουν τους καρπούς της προσπάθειας να συμφωνήσουν με το Συμβουλίο και στο μέλλον. Όσον αφορά ακριβώς αυτές τις ε, συνδεδεμένες ενισχύσεις, για μένα είναι απόλυτη προτεραιότητα ε, στη Γαλλία που είναι μεγάλη χώρα υπάρχουν και μεγάλη ποικιλία καταστάσεων οπότε χρειάζεται να μείνουν αυτά τα μέτρα για όποιον έχει προβλήματα ε, εκεί που έχουμε κτηνοτροφία σε χορτολιβαδικές εκτάσεις κυρία Ρανσνέ ναι, μας λέτε για τις 150.000 ευρώ ε, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει κάποιο είδους τέλος, κάποιο είδους επιβάρυνση για να, χρημα... για να χρηματοδοτηθούν οι γεωργοί. Όμως προσοχή, γιατί στην προηγούμενη κάπου αυτό δεν υλοποιήθηκε. Από την κατάρριξη των πρώτων εκταρίων. Να προσέξουμε αυτό το μέτρο. Έτσι βοηθούνται οι μικροεκμεταλλεύσεις. Και όσον αφορά τον πελοενικό τομέα έχουμε τις προτάσεις της Επιτροπής για να υπάρχει άνω όριο συνισχύσεις. Προσοχή να μην ξεπεράσουμε αυτό το άνω όριο γιατί έτσι θα προσκάψουμε, θα στρεβλώσουμε την αγορά. Ο επόμενος, ο, ο κύριος Μπούντα, μπράβο στους οι ηγητές και στην εισηγητρία βέβαια θέλω να πω τα εξής. Πρώτον, σύγκληση Είπαμε ότι θέλουμε ένα αποτελεσματική ΚΑΠ σε σχέση με όλους τους ε, γεωργούς. Αλλά αυτό σημαίνει και σε Ανατολή και Δύση να έχουμε τις ε, ίδιες πληρωμές και ενισχύσεις. Όμως δεν μπορούμε να έχουμε ίσους όλους το παιχνίδι γιατί ε, υπάρχει μεγάλη ανισότητα στις επιδοτήσεις, στις ενισχύσεις. Πώς θα έχουμε επομένως τη σύγκληση τώρα για τους νέους ερχόμενους στην Γεωργία. Πρόκειται για μια κατηγορία γεωργών. Πολλές φορές ε, αυτοί είναι νέοι, αλλά δεν αρκεί αυτό για να καλύψουμε την απερίμωση της ε, υπαίθρου. Άρα να τους βοηθήσουμε αυτούς τους νέους ερχομένους. Τώρα όσον αφορά το ανώριο, το κάπινγκ, τα συζητήσαμε με τους Ρουμάνους Γιώργους και οι μεγαλοκαλλιεργητές έχουν δανειστεί, έχουν κάποιο στεγαστικό για να πάρουν το δάνειο για την εκμετάλλευση και έχουν υποβάλει στην τράπεζα τις επιδοτήσεις που παίρνουν. Αλλά αν δεν τους δώσουμε την ε, επιδότηση, πάει η περιουσία τους. Δεν μπορούν να καλύψουν την δανειοδότηση. Συμφωνώ με τον κύριο Ντόρφμαν. Ε, βέβαια στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχουν και κάποιες ε, απάτες, κάποιο είδου κερδοσκοπία, αλλά υπάρχουν και οι καλόπιστοι, αυτοί που βάλανε υποθήκη το σπίτι τους. Αυτοί θα χάσουν τη γη τους, θα χρεοκοπήσουν. Να το έχουμε αυτό βάρος στη συνείδησή μας. Μα ποιος θα μπορέσει να ισχυριστεί στους φόρους του ότι ένα τέτοιο μέτρο είναι θετικό. Επίσης επιμένω, θα πρέπει να μην υπάρχει η προϋπόθεση της ταυτοποίησης των ζώων γιατί έτσι τιμωρούμε αθώους. Κολομπιέ. Βέβαια, να μην αμφισβητήσουμε αυτά τα οποία έγινε, ιδίω όσον αφορά τα υπέρ των μικρομεσαίων ε, εκμεταλλεύσεων. Όμως είναι επικίνδυνο ε, όλα αυτά να, δημοσιονομικά να τα κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται να δούμε η μεταρρύθμιση, πώς δεν θα επιβληθεί ε, δια της βίας με, μαζί με ένα δημοσιονομικό ναυάγιο. Θα πρέπει, από ό,τι από την Επιτροπή, ότι θα πρέπει να ισχύσει ότι ισχύει για έλεγχο και πιστοποίηση. Αλλά τι θα ελέγξουμε και τι θα πιστοποιούμε. Τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε ε, σωστή αντίληψη για τη μεσονομική κάλυψη της μέλους σας ΚΑΠ. Το άκουσα από τους συναδέλφους. Και αυτά τα λέω και τα ξαναλέω σε όλες τις επιτροπές και για τους νέους γεωργούς, σχεδόν ένας στους δύο. Ε, δεν καλύπτεται από τις ενισχύσεις και αυτό δεν να μας προβληματίσει. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Έρενς Καρδία ακόμα και αν δεν πρόφερα καλά το όνομά της. Λέω μιλήτρια η κυρία Ριμπέιρο. Δεν είναι δυνατόν να μειωθούν τα τα όρια για μένα. Οι άκρος απόμακρες περιφέρειες θα υποφέρουν από κάτι τέτοιο. Θα δυσκολευτούν πολύ. Επίσης βλέπουμε ότι Όσον αφορά τη δομή του δεύτερου πυλώνα για τις άκρος απόμακρες περιφέρειες, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Έχουμε αυτονομία, έχουμε κυβέρνηση και κοινοβούλιο ως αυτόνομη περιφέρεια. Και δεν είναι δυνατόν να εξαρτώμεθα από την κεντρική κυβέρνηση η οποία θα μας βάζει εμπόδια στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Έπειτα, για τα άλλα προγράμματα. Ξέρω ότι τα στηρίζει η συγγήτρια και μπράβο της, αλλά έχουμε ένα σύστημα τώρα που δημιουργεί κάποιο κενό, γιατί βάζει τις απόμακρες περιφέρειες στην ίδια μοίρα με τις περιφέρειες στην υπηρετική χώρα. Θα έπρεπε να υπάρχει διαπραγμάτευση συγκεκριμένα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άκρος απόμακρες περιφέρειες. Αυτές τις ιδιαιτερότητες πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας και συγγνώμη που κακοποίησα το όνομά σας στην αρχή, κυρία Ρέντς. Ευχαριστούμε. Επόμενος, ο κύριος Λουαζό. Για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι ποσά θα δεσμευτούν σε αυτήν τη νέα κοινή γεωργική πολιτική. Εννοείται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να δεχτεί μείωση του προπολογισμού και πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να αλλάξουμε την πρόταση στην περίπτωση που δεν μας ικανομήσει το πλαίσιο. Νομίζω ότι συμφωνούμε, κύριε Συγκήτρια, γι' αυτό. Πολύ λιγότερο όμω με το γενικό πνεύμα τη έκθεσή σα. Πρώτα απ' όλα, βάζετε σαν στόχο να αποφύγουμε κάθε κίνδυνο επανεθνικοποίηση τη ΚΑΠ. Μα αν λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες όλων των περιφερειών, μόνο τότε θα καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα σε κάθε χώρα μέλος χωριστά. Ναι, είναι μεγάλα λόγια αυτά, όχι στην επανεθνικοποίηση. Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι διάφοροι τομείς θα ενισχύονταν σε εθνικό επίπεδο πριν βρεθούν εκτεθειμένοι στους ε, κανόνες και τον ανταγωνισμό της αγοράς που είναι πάντα ακραίοι. οι κανόνες που είναι πάρα πολλοί, έχει σαν αποτέλεσμα τώρα να πρέπει να αποφασίσει ο συνομοθέτης και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο επίσης λειτουργίας και στο τι παραχωρούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας ώστε οι αγρότες να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Γιατί να μην στηρίξουμε τα μέτρα παρέμβαση στην αγορά. Και γιατί να μην καταγγείλουμε την εμπορική πολιτική στα γεωργικά προϊόντα. Γιατί να μην θέσουμε υπό το δόγμα των ελεύθερων συναλλαγών που τόσο πολύ πλήττει τη γεωργία μας. Και όσον αφορά το περιβάλλον, πιστεύετε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την αιρεσιμότητα με τις κυρώσεις για να καταλήξουμε σε μια πολιτική με κίνητρα που να επιβραβεύει τους αγρότες που προστατεύουν το περιβάλλον θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα κείμενο που να προσφέρει εγγύηση στον αγρότη από διάφορους κινδύνους, διακόπτει ο πρόεδρος. Ο κύριος Γιάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι δεν θα διαρκέσει για πάντα η γη στον πλανήτη, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε ακόμα 6.000 χρόνια έχουν υπολογίσει. Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν το μέλλον τη γεωργική πολιτική, γιατί υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που φαίνεται ότι θέλουν να κάνουν πολιτική αυτοκτονία. Εμεί είμαστε όμω πολιτικοί και οι πολιτικοί, οι επαγγελματίε πολιτικοί, καταλήγουν στου συμβιβασμού. Αυτή είναι η άποψη τη ομάδα μου. Προσπαθούμε να βρούμε λοιπόν συμβιβασμού και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Έχουμε ένα από, παράδειγμα, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ε, σταδιακή μείωση και τα κάπινγκ. Αυτό που περιέγραψε ο κύριος εγώ ούτε αυτό μου αρέσει, αλλά θα γίνει κάποια έρευνα για το πώς μπορούμε να το αποφύγουμε. Ένα παράδειγμα. Έχουμε δύο οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν θέλουμε να τις τιμωρήσουμε. Γιατί θέλουν να έχουν ε, τακτικές ε, ε, ώρες εργασίας ε, ή για παράδειγμα ε, τακτικές διακοπές. Πάντα δηλαδή εξορισμού η πιο μεγάλη έκταση είναι χειρότερη. Δεν είμαι σίγουρος. Θα πρέπει να προσέξουμε στη τελική ανάλυση πάντα στο επίκεντρο να είναι ο αγρότης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους απογραφειοκρατικοποίησης θα πρέπει σε ό,τι αφορά τα θέματα ρεσιμότητας, σε ό,τι αφορά τα θέματα της υπερεκμετάλλευσης των ε, επιφανειών, να δούμε ένα ποσό κατά αποκοπή και το καθεξό, καθεξής. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν με τις νέες προτάσεις να παραμείνει βιώσιμη και η πολιτική, η γεωργική. Και εδώ θέλουμε να κοιτάξουμε και τα εθνικά σχέδια, να δούμε ποιε είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι υπέρ των ε, οικοσκήμ, των οικολογικών αυτών πολιτικών και πιστεύω ότι θα πρέπει να βγουν στην δεύτερη ε, πυλώνα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Πρόεδρε, λέει η κυρία Σέντερ Ροντρίγκε, θέλω να θίξω δύο-τρία ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, τα νότια τόρια είναι πάρα πολύ βασικά. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε, να εφαρμόσουμε τα νότατα όρια στις ενισχύσεις, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να κατανείμουμε τα ποσά και να ενισχύσουμε την μικρή και μεσαία καλλιέργεια. Εμείς προτείναμε, ή εγώ πρότεινα με τις τροπολογίες μου, τριών ειδών ανώτατα όρια, ένα 30.000 ευρώ, για κάθε εκμετάλλευση σε μη ευνοημένες περιοχές, 50.000 για τις κανονικές και 60.000 στις ορεινές ε, περιφέρειες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι ένας τρόπος να ανακατανύμουμε τα ποσά και να στηρίξουμε την μικρή και μεσαία γεωργία, γεωργική εκμετάλλευση. Τώρα, μιλάμε για μια πολιτική που δεν θέλουμε να έχει την τιμή στο κέντρο της συζήτησης. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει ενίσχυση για τους αγρότες, άντρες και γυναίκες των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων Ο κύριο στοιχείο μια σημαντική ενίσχυση η οποία να τους επιτρέπει να επιβιώνουν. Πέρα από τις ενισχύσεις από άλλες πηγές. Είναι πολύ βασικό, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στις συζητήσεις μας. Θέλουμε να διατηρήσουμε τους ανθρώπους στις γεωργικές περιοχές, να παράγουν προϊόντα και όχι να εγκαταλείψουν την γεωργική δραστηριότητα. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι πολύ καλός ορισμός του τι είναι πραγματικός αγρότης. Πλήρους απασχόλησης και μερικής απασχόλησης. Μόνο αυτοί θα έπρεπε να παίρνουν ενισχύσεις. Τέλος, και εγώ θα ήθελα να γνωρίζω γιατί ο Επίτροπος συνέχεια ρωτάει πότε θα ψηφίσουμε την ΚΑΠ. Μα τι γίνεται. Δεν θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει το χρόνο που χρειάζεται για να κάνει καλά τη δουλειά του. Τι είναι αυτή η εκβιασμή από την Επιτροπή πότε και πότε. Η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την κυρία Χεράνς Καρθία, για τον κόπο που έχει κάνει και για τον χρόνο που έχει αφιερώσει σε αυτό το περίπλοκο θέμα. Θέλω πραγματικά να τη συγχαρώ, γιατί βρήκε αρκετό χρόνο για να ακούσει και τους εκπροσώπους όλων των χωρών μελών και για να λάβει η υπόψη της τις θέσεις μας, τις διαφορές μας και να προσπαθήσει να καταλήξει σε συμβαστικές τροπολογίες προκειμένου η κοινή γεωργική πολιτική να διατηρηθεί ευρωπαϊκή, ενώ συγχρόνως δίνουμε στο καθένα τη δυνατότητα να βρει τα πράγματα που τον εξυπηρετούν καλύτερα. Θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία οι νέοι αγρότες. Βλέπω ότι συμφωνούμε με αυτό όλοι και η συγκίτρια στηρίζει τις δικές μας προτάσεις. Θα μας στηρίξει και η Επιτροπή. Πιστεύω. Αυτό που θέλω κυρίως να τονίσω είναι τη θέση των γυναικών στην Ήπεθρο. Μέχρι τώρα οι γυναίκες ήταν αόρατες στην Ήπαθρο. Έχω καταθέσει πολλές τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και η κυρία Έρενς Καρθία ε, τις έλαβε υπόψη της γιατί θέλει να βοηθήσει τις γυναίκες που ζουν στην Ήπεθρο και να υποστηρίξει προγράμματα υπέρ των γυναικών αυτών. Δυστυχώς όμως η Επιτροπή βλέπω ότι θέλει να τα αφαιρέσει αυτά. Εγώ δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό. Μέσα από αυτή τη συζήτηση λοιπόν θέλω να στηρίξω και πάλι χωρίς καμία επιφύλαξη θα πρέπει όλοι να βρούμε την καλύτερη ε, λύση για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Αντρία. Ομολογώ ότι είμαι ανήσυχο από τη συζήτηση που παρακολουθώ. Γιατί η συζήτηση γίνεται ε, σαν να συζητούσαμε για μία έκθεση πρωτοβουλίας ή μόλις αρχίσαμε να συζητάμε για τη νέα κοινή γεωργική πολιτική. Είμαστε όμως ε, στις 29 Ιανουαρίου και γύρω στις 6 Φεβρουαρίου πρέπει να ψηφίσουμε. Ε, δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Και από αυτά που ακούω στη συζήτηση βλέπω ότι κάθε άλλο παρακοντά στη λύση είμαστε. Το σχέδιο μεταρρύθμισης, το οποίο εμεί ποτέ δεν είδαμε σαν ένα πραγματικό σχέδιο μεταρρύθμισης, λίγο πολύ μας είπαν ότι πρόκειται για τεχνικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Ενώ διαπιστώνουμε από τη συζήτηση ότι ούτε απλοποίηση έχουμε, ούτε έχουν λυθεί τα προβλήματα. Ανησυχώ λοιπόν με το χρονοδιάγραμμα αυτό που έχουμε μπροστά μας. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταλάβει ότι όταν έχουμε δύο συνομοθέτες, αυτό πετύχει χρόνο για να κάνουμε καλά τη δουλειά μας ως ευρωβουλευτές. Αυτά τα πηγενέλα με τους διάφορους τομείς δεν μας οδηγεί σε λύση θα πρέπει να μπούμε περισσότερο σε βάθος για πολλά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα σε τρία. Το ανώτατο όριο είναι ζωτική σημασία και για μένα, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο, ακόμα και αν είναι υψηλό το ανώτατο όριο. Πρέπει όμως να συνδέεται και με τις ε, αναδιαναμητικές ενισχύσεις επίσης. Αν υπάρχει απασχόληση, είναι καλό να υπάρχει αυτή η αναδιανεμητική ενίσχυση. Και το θέμα της ε, σύνδεσης είναι κάτι που πρέπει να διευκρινίσουμε περισσότερο. Τελείως. Δεν θα ήταν υπεύθυνο από την πλευρά μας να φτάσουμε σε τριμερή διάλογο έχοντας μια αδύναμη θέση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα έπρεπε. Θα το μετανιώσουμε στο μέλλον σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θυμάμαι ότι 15 χρόνια δουλεύουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τότε που ήρθα εγώ και ξέρω ότι ποτέ δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε αρκετά αυτά που θέλαμε. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, εκπρόσωπο της Επιτροπής και εγώ να συγχαρώ τους και και την συγγητρία για τη δουλειά τους για να μπορέσουν τις 5.500 περίπου τροπολογίες να τις κάνουν κάτι πιο λογικό και έτσι με τον τριμερή διάλογο να έχουμε καλή ε, χειρισμούς. Ό,τι τεχνική βοήθεια μπορούμε να δώσουμε, ευχαρίστως να σας βοηθήσουμε έτσι και να κινηθούμε μέσα στις προθεσμίες. περιορίζουμε σε κάποιο για γενικόλογα θέματα και μετά θα σας πω για δύο-τρία συγκεκριμένα. Πρώτα-πρώτα υπενθυμίζω ότι το νέο μοντέλο το οποίο προτείνουμε δεν συνεπάγεται ότι το παρόν σύστημα της συμμόρφωσης που έχει να κάνει με τους ουσιαστικούς και τον οριζόντιο κανονισμό θα φύγει και είναι μόνο το ένα η μία μία όψη του τους. αυτο Αυτό πάει χέρι-χέρι με την επικουρικότητα. Θα καλύψουμε ό,τι χρειάζεται κάθε κράτο μέλος, άρα πρέπει να του αφήσουμε κάποια περιθώρια και ό,τι κοινοί κανόνες θεσπιστούν θα περιορίζονται στα βασικά. Σε ό,τι θεωρούμε αναγκαίο τόσο ώστε η πολιτική μας είναι πραγματικά κοινή. Γι' αυτό με τις προτάσεις μας θελήσαμε να έχουμε παρεμβάσεις μόνο στις άμεσες πληρωμές, στα προγράμματα, το ελάχιστο δηλαδή. Και καλό με τα κρατη θα κάνουν ό,τι θέλουν για τις ειδικότερε ανάγκες τους. Διαπραγματεύσεις θα γίνουν, όπου θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά να μην διαλύσουμε το σύστημα με τις διαπραγματεύσεις. Να μην επιστρέψουμε στο σημείο που τα κράτη-μέλη να λένε θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό για τους γεωργούς, για το περιβάλλον, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί μας περιορίζουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν δύο χρόνια για να εφαρμοστούν οι αλλαγές τους. Μην πάμε λοιπόν σε τέτοιο καθεστώς λεπτομερών ρυθμίσεων. Το είπατε μερικοί από σήμερα. Πάμε επομένω έτσι στο παλιό σύστημα των ελέγχων και των χρόνων ελέγχων. Δεν το θέλουμε αυτό, να το θέλουμε το αντικαταστήσουμε για σύστημα ελαφρότερο επί τη βάση τη επίδοσης αυτά που είπαμε νωρίτερα σήμερα. Συγκεκριμένα παραδείγματα πολλοί από εσά ανέφεραν τις πάγιε μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις ρυθμίσαμε τη μεταρρύθμιση του 2013 και καλύψαμε το πλήμα των κρατών μελών για αυτές τις εκτάσεις με τις διαπραγματεύσεις του Omnibus που ολοκληρώθηκαν το 2017 τώρα. Τι προτείνουμε. Μείωση του ελάχιστου αυτών των εκτάσεων με τις ελάχιστες κοινές ρυθμίσεις για όλα τα κρατημέλη. Ήδη έχουν ευελιξία τα κρατημέλη όσον αφορά τον ορισμό αυτών των χορτολιβαδικών εκτάσεων. Οπότε, είπαμε ότι αυτοί οι ορισμοί, αυτά που προβλέπονται ήδη, να τα κάνουν ό,τι θέλουν στα πλαίσια των αναγκών του στα κράτη-μέλη. Τώρα, ο ορισμός του Γιώργου που έχουμε τώρα ήταν ένα βάρος για κράτη-μέλη και έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα στο ζήγισμα κόστους ωφέλους. Θέλουν τα κρατημέλια. να έχουν ελέγχους ούτω ώστε να υπάρχει έλεγχο στο ποιο παίρνει τι ενισχύσει. Γι' αυτό εμεί είπαμε να είναι εκουσίου χαρακτήρα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει στοχοθέτηση αυτών των ελέγχων. Αυτό είναι το πνεύμα των ε, προτασιών μας όσον αφορά τον ορισμό του πραγματικού αγρότη. Άλλο. Είπαμε ότι από το σύστημα της συμμόρφωσης πάμε σε σύστημα επιδόσεων. Οπότε θα πρέπει το νέο σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Τι χρειάζεται. Θα πρέπει να επιτρέψει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρεί τις δεσμεύσεις της για την ετήσια απαλλαγή που χορηγεί το Κοινοβούλιο. Άρα χρειάζονται ετήσια στοιχεία, όπως και σήμερα. Αλλά αυτό όσον αφορά τις επιδόσεις και όχι την συμμόρφωση. Άρα χρειάζονται εκθέσεις των κρατών μελών στην Επιτροπή. Και μας χρειάζεται και για την ετήσια απαλλαγή. Να πάμε σε σύστημα αναδιετίας, ε, έκθεσης ε, κάποιο μεσοπρόθεσμο σύστημα αξιολόγησης. Α, αυτό θα ήταν ένα πλήγμα στο σύστημα. Δεν θα λειτουργούσε πια. Θυμηθείτε το αυτό. Όταν συζητήσουμε τα επιμέρους της πρότασής μας. Όσον αφορά προγράμματα και εκθέσεις κρατών μελών. Πάμε τώρα στο θέμα των προθεσμιών, Τις προθεσμίες. 15 Δευτέρου όσον αφορά τις εκθέσεις των επιδόσεων. Ετήσιε εκθέσει Μερικοί ανησυχούν. Δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να το τηρήσουν. Θέλουν πιο πολύ χρόνο να μαζέψουν τα στοιχεία που ζητούμε εμείς για αυτές τι εκθέσει Τι λέμε. Όσοι επιδοπλίστων θα αναφέρουν ποσοτικά στοιχεία μέσω του συστήματος πληροφορικής. 75-80% αφορούν κάποια μέτρα, κάποιες παρεμβάσεις και για τις οποίες θα πρέπει να έχουν δοθεί μέχρι 30 Ιουνίου και οπότε κατόπιν έχουμε τα στοιχεία στους οργανισμούς πληρωμών του κράτους μέλους και μετά έχουν το υπόλοιπο της χρονιάς για να κάνουν την έκθεση. Και αυτές οι εκθέσεις ως πονδυλική στήλη έχουν τους output indicators και από την άλλη μεριά έχουν τους result indicators. Output indicators είναι κάποιες πληροφορίες ποσοτικές όπως ο αριθμός των εκταρίων. Αυτά υπάρχουν ε, στο σύστημα πληροφορίων των μελών. Δεν είναι καμιά πυρηνική φυσική, εύκολο να τα μαζέψουν τα κράτη. Και result indicators είναι η απόκληση από την προηγούμενη χρονιά, η ποσοτική αύξηση δηλαδή. νεκτάρια βιολογική παραγωγή, από το τέλος χρονιάς μέχρι την, ε, την, το συν 1. Και έτσι υπολογίζει Η διαφορά στο ποσοστό και το λέτε στην Κομισιόν. Έτσι είναι διαχειρίσιμο, έτσι λειτουργεί το σύστημα με αυτές τις ενέργειες ετησίως συγκεκριμένα θέματα τώρα. Στόχοι. Είναι οι στόχοι στην καρδιά του της πρότασής Είπατε να αλλάξει η διατύπωση. Προσοχή όμως, όταν αλλάζουμε τη διατύπωση των στόχων, των νέων στόχων, να ξέρουμε ότι αυτό έχει επιπτώσεις και στους δείκτες οι οποίοι είναι στο παράρτημα 1 της πρότασης όπου λέει για την έκθεση κράτους μέλους. Άρα, αν αλλάξει το ένα, θα αλλάξει και το άλλο για να ταιριάζουμε το σύστημα. Δεύτερο σημείο για τις εφαρμοστικές κατεξοδόσεις πράξεις. Είπατε ότι παραέχουμε πολλές τέτοιες. Για καθίστε και δείτε τι προβλέπετε στους σημερινούς κανονισμούς και συγκρίνεται τέτοιες πράξεις που έχουν οι τωρινοί κανονισμοί. Οι δύο τωρινοί κανονισμοί, οριζόντιος και αυτός για τα στρατηγικά προγράμματα. Η μισή είναι τώρα. Τους μισούς προβλέπουν οι τωρινές προτάσεις. Άρα μην το πειράξετε. Αυτό το σημείο. Κάτι άλλο επίσης το οποίο έχει πολιτικό χαρακτήρα, έχει σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις διαπραγματεύσεις. Οι αναδυναμητικές πληρωμές και το κάπινγκ σύμφωνα με προτάσεις μας έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα ούτω ώστε να στοχεύσουμε τις πληρωμές, να βοηθήσουν τους μικρό γεωργούς, μικρό καλλιεργητές. Όχι. Θα πρέπει αυτά χέρι-χέρι να υλοποιηθούν από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Τώρα για τις εξόχως μακρινές περιφερειακές περιφέρειες, ευελιξία και ελευθερία για τα κράτη-μέλη να κάνουν τα στρατηγικά τους προγράμματα. Αυτά τα κράτη που έχουν τέτοιες περιφέρειες μπορούν να ρυθμίσουν τα πράγματα σύμφωνα με τις ιδιομορφίες αυτών των περιφερειών ή περιοχών. Η περιοχων πολύ. Πρώτα απ' όλα, όλους σας ευχαριστώ πραγματικά για τα σχόλιά σας και για τη συνεργασία σας. Όντως είναι περίπλοκο το θέμα και γι' αυτό Ευχαριστώ για τη στήριξή σας και εν ώψη μάλιστα των ευρωεκλογών και βέβαια αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει και μετά. Είναι και ένα θέμα που απασχολεί πολύ και τα μέσα ενημέρωσης. Είναι λογικό να γίνονται πολλές συζητήσεις και να υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις, γιατί εκπροσωπούμε όλο το ιδεολογικό φάσμα. Τελειώνει και η θητεία, όλοι είμαστε πιο εκνευρισμένοι, τι να κάνουμε. Για τη μεθοδολογία. Ε, μου κάνει εντύπωση που με ρωτάτε γι' αυτό. Για τη μεθοδολογία σε κάθε νομοθετική έκθεση ίδια είναι. Συγκεντρώνονται οι πρωτολογίε από τον εισηγητή, οργανώνονται, εξετάζονται, τοποθετεί το εισηγητή και εκπονεί πρόταση, η οποία να συμπεριλαμβάνει όσο γίνεται ε, περισσότερε από τι τοποθετήσει που εκφράζονται με τι τροπολογίε. Μετά γίνεται συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο και μετά όπου υπάρχουν πολεμικά σημεία ή που στα τεχνικά δεν μπορούμε να συζητήσουμε, πάμε στους σκιώδεις και εκεί αποφασίζουμε είτε με ομοφωνία, τόσο το καλύτερο, ή με πλειοψηφία, συνήθως με πλειοψηφία. Άρθρο, άρθρο, ναι βεβαίως, άρθρο, άρθρο. Πολλές φορές οι συζητήσεις γίνονται για μία λέξη, για ένα επίθετο, για ένα άρθρο, για ένα πολύ μικρό κομματάκι της πρότασης μπορεί να συζητήσουμε για πολύ καιρό. Οπότε, φυσικά και εξετάζουμε άρθρο-άρθρο. Γιατί θέλουμε να ξέρουμε αν τελικά θέλουμε να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά, αν συμφωνούμε ή όχι. Ναι, Μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε μια τεχνική συνάντηση και μετά να πάμε σε μια άλλη και μετά σε σκιώδες. Μπορεί να ξανανοίξει η συζήτηση γιατί κάποιος στην τελευταία συνάντηση προτείνει ένα νέο άρθρο, μια νέα λέξη και ξανασυζητιέται το θέμα και αυτού και από την αρχή. Χάος λοιπόν. Χάος επειδή γίνονται προτάσεις μαξιμαλιστικές και ο καθένα πιστεύει ότι η δικιά του η πρόταση είναι καλύτερη και η δικιά του είναι η απόλυτη αλήθεια. Χάος, γιατί όλοι θέλουν το δικό τους και δεν δίνουν σημασία στο τι λένε οι υπόλοιποι. Τρεις και συζητητέ για κάθε έγγραφο. Χάς να φτάνουμε σε μια τεχνική συνέντηση και μια πολιτική ομάδα να έχετε με πέντε ανθρώπους ή να είμαστε και κλεισμένο το θυρών και να κάθεται κάποιο και να μιλάει σε Skype με κάποιους που να παίξω. Ε, τι και κλεισμένο το θυρών τότε. Έτσι είναι το χάο. Γι' αυτό έχουμε χάο. Λοιπόν, άκουσα την κυρία Αγγιλέρα, Αγγιλέρα έφυγε δυστυχώ κρίμα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τελικά η θέση που γνωρίζουμε ότι υποστηρίζει η ομάδα τη δεν είναι αυτή που μα παρουσίασε εκείνη. Δεν ξέρω οι σοσιαλιστέ πόσε φορέ συνεδρίασαν ή πώ είναι οργανωμένοι και αν κάνουν το ίδιο και άλλες πολιτικές ομάδες, αλλά θα έλεγα ότι στο ΕΛΚ συνεδριάζουμε κάθε τόσο, είμαστε στην πέμπτη συνάντηση και όταν έχουμε μια τοποθέτηση πάμε παραπέρα. Τη λέμε και σε ολόκληρη την ομάδα. Η συζήτηση, ναι, γίνεται στη γλώσσα του Σέξπιρ, όπω είπατε σωστά, στα αγγλικά, όταν είμαστε μεταξύ μα, τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε ένα τον άλλον και να προχωρήσουμε. Η κυρία Νόχελ ούτε και αυτή είναι εδώ. Κρίμα. Θα ήθελα να είναι εδώ. Να οργανωθούν. Πρέπει να οργανωθούν. Τι να κάνουμε. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν ως μεταπολιτικοί να απορρίπτουν την διαπραγμάτευση σε ό,τι και αν καταλήξουμε με τις σεβαστικές τροπολογίες. Ε, ας το λέγανε νωρίτερα τουλάχιστον. Γιατί όποιος δεν θέλει να πετύχει μια διαπραγμάτευση, γιατί δεν θέλει συμφωνία, ε, να μας το λένε από πριν. Και να μαζευόμαστε οι υπόλοιποι που θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, που θέλουν να είναι επικοδομητικοί στις διαπραγματεύσεις και να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα και αποτέλεσμα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ο κύριος Βάης με ρώτησε για ποιος είναι ο πραγματικός ε, αγρότης. Η πρότασή μου είναι σαφής. Ποια είναι η δικιά μου ιδέα δηλαδή για το ποιος είναι πραγματικός αγρότης. Υπήρξε πρόταση συμβιβαστική για το ποιος είναι πραγματικός αγρότης και Θυμίζει πολύ την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρί να είναι ακριβώ το ίδιο, γιατί αφήνει ευελιξία στι χώρε μέλη. Και ξέρετε γιατί. Γιατί στη Ρουμανία, για παράδειγμα, από ό,τι άκουσα από συναδέρφου μου στην κοινοβουλευτική μου ομάδα, έχουν πρόβλημα. Δεν μπορούν να ζήσουν μόνο από τη γεωργία. Οι περισσότεροι αγρότες έχουν και δεύτερο επάγγελμα, οπότε πρέπει να αφήνουμε ελευθερία στις χώρες μέλη για να προσαρμόσουν τον ορισμό στη δικιά τους πραγματικότητα. Μου φαίνεται πιο λογικό αυτό. Αλλιώς είναι σαν να πηγαίνουμε με το κεφάλι στον τοίχο για να σπάσουμε το κεφάλι μας. Αυτός ο ορισμός μάλιστα συνδέει την παραγωγική δραστηριότητα με τον ορισμό. Ξέρω ότι δεν της αρέσει η σύνδεση αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί λέω ότι θα έχουμε προβλήματα στον ΠΟΕ. Επίσης, και υπόθεκε γι' αυτό, πρέπει να διατηρήσουμε και την οικογενειακή γεωργία και να την υποστηρίξουμε. Ο κύριος Νταντά μου υπενθύμησε τη συμφωνία Omnibus και έχει δίκιο γιατί κρίθηκαν πριν από ένα χρόνο, 13 μήνες και βοήθησαν να λυθούν πολλά προβλήματα. Αν συμφωνήσουμε σε κάτι που το βελτιώνει, το καλύτερο. Αλλιώς να παραμείνουμε σε αυτό. Και αυτό λένε με τις τροπολογίες τους πολλοί να επιστρέψουμε στο όμνιμπους. Αν καταλήξουμε σε ομοφωνία όλοι, το στο καλύτερο η πλειοψηφία, εντάξει. Αλλιώς έχουμε ήδη ένα καλό έγγραφο για να μείνουμε σε αυτό. Αναφερθήκατε σε αυτούς που εγκαθίστανται ως νέοι αγρότες ανεξαρτήτως ηλικίας. Χρειάζονται, είναι μια πραγματικότητα σε πολλές χώρες. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είτε για πρώτη φορά μπαίνουν στον τομέα, ή επιστρέφουν γιατί διέκοψαν την γεωργική τους δραστηριότητα, αλλά επιστρέφουν. Τέλος, ε, κύριε Αντρέου, η συνδεδεμένη ενίσχυση την Όταν δραστηριοτητα στις ομάδες αυτή η πρόταση, πήγε και στο σκιώδη σας συζητητή. Εγώ είμαι ανοιχτή τεχνικά. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ. και επιτελεστεί πρόοδος αλλά και στο ΕΛΚ συζητάμε ξανά και ξανά. Φαντάζομαι και οι υπόλοιπε ομάδε και ελπίζω να καταλήγουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να συμφωνήσω και να ευχαριστήσω και εγώ την ε, εισηγήτρια τη γραμματεία, το προσωπικό και νομίζω ότι παρά τις διαφορές μας προχωράμε. Και να έχουμε υπόψη μας ότι έχουμε πετύχει και τώρα. Σας ευχαριστώ και πάλι και τώρα προχωράμε. στον κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς και τον ε, εισηγητή μας, ο κ. Ανδρέα. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, je voudrais, si vous me permettez, juste avoir un propos euh, liminaire sur, sur la dette. Θα είμαι συνοπτικός. Θέλω να πω κάτι για τα όσα ακούσαμε τώρα για την κυρία Νότον Καρθία. Μπράβο, μπράβο για τη δουλειά της. Κάτι πολύ συγκεκριμένο. είναι συμπαγές το ΕΛΚ. Έχουμε τις ε, τροπολογίες του συντονιστή που αφορά αυτή την πρόταση της μεταρρύθμισης. Η περίπλοκη είναι πάντως κατάσταση και στη δική του ομάδα και στη δική μας. Πάντως, να ευχαριστήσουμε την γραμματεία της Επιτροπής μας τους βοηθούς μας, των πολιτικών ομάδων, τους βοηθούς μας, όλους τους αδελφούς, γιατί είναι τόσο δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβασμό για τόσο δύσκολο θέμα. Αυτό το σύστημα τώρα το επεξεργαζόμαστε, το εξειδικεύουμε. Έχουμε δικές διατάξεις για το Αιγαίο, τη, τις ε, περιφέρειες τις απότερες και έχουμε όλες αυτές τις τροπολογίες 94 τις οποίες αφορούν την οτιολογική έκθεση και μένουν άλλες 500 τόσες για την τροποποίηση του κανονισμού. Έχουμε ήδη τέσσερις συναντήσεις και άλλες δύο μέσα στο Φεβρουάριο, με το τέλος Φεβρουάριο. Ήδη κάναμε τρεις συναντήσεις. Οι σκιώδες ηγητές και ένα σωρό τροπολογίες ήδη τις έχουμε συζητήσει, σκιώδες και φτάσαμε τις 400 και οπότε με όλα αυτά τώρα πάμε για συμβαστικές τροπολογίες μέχρι σήμερα. Επομένως αυτά πετύχαμε. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τα μεταλλαγμένα. Σχεδόν έχει κλείσει το θέμα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή του πρώτου άρθρου σε σχέση με τις ε, χρηματαγορές και για την παρέμβαση. Αυτά που λέει το άρθρο 3. Συμφωνήσαμε και οι και όσον αφορά τη θέση σε εμπορία του άρθρου 6 επίσης συμφωνούμε. Επίσης όσον αφορά κατόφλι αναφοράς του άρθρου 7 συμφωνούμε. Αλλά το δικαστήριο διέγραψε ακύρωσε αυτό το άρθρο επίσης και για το άρθρο 11 έχουμε συμφωνήσει για την περίοδο της κρατικής παρέμβασης που είναι το άρθρο 12 συμφωνήσαμε και για το χρονικό πλαίσιο του άρθρου 13. Όσον αφορά τα αμπελοϊνικά έχουμε το άρθρο 61. Συμφωνήσαμε τότε την ανταλλαγή απόψεων, η ανταλλαγή ή οι και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προστασία των ονοματών προέλευσης είναι το άρθρο 96 τρόσον αφορά της κατεξούδας πράξεις για τα αμπελοϊνικά προβλέπονται αυτά στο βασικό κανονισμό και εδώ συμφωνήσαμε ισχυώδης. Για όλα αυτά που καλύψαμε και έχουν συμφωνηθεί για διάφορες περιφέρειες θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το άρθρο 14 για τον καταλογισμό αλλά υπάρχει πρόβλημα διατύπωσης οπότε θα πρέπει να το ξαναδούμε αλλά δεν υπάρχει διαφωνία επί της ουσίας και επίσης η κρατική επανέβαση του άρθρου 15 θα πρέπει να το ξαναδούμε για να χτενίσουμε την διατύπωση δεν υπάρχει πολιτικό πρόβλημα. Κατανάλωση στα σχολεία λαχανικών και φρούτων. Εκεί έγινε εκτενή συζήτηση και συμφωνούμε για την ε, ε, κάλυψη αυτού του θέματος από το στρατηγικό πρόγραμμα. Ξεργαζόμαστε μία διάταξη ή μία τροπολογία συμβαστική Τώρα, επίσης για τα αμπελοενικά, για τον μηχανισμό διαφύλαξης του άρθρου 63 και αυτό συζητείται σε τεχνικό επίπεδο για να δούμε εκεί τι ορισμό εκμετάλλευση θα δούμε. Τώρα 70, 64. Και εδώ το συζητούμε τώρα για τις οργανώσεις παραγωγών. Δεν το συζητήσαμε αλλά συζητείται από τη τεχνική ομάδα. Για τα παραρτήματα έχουμε την κοινή οργάνωση αγοράς και σήμερα τα συζητήσαμε όσον αφορά το κρασί χωρίς νόπνευμα συμφωνήσαμε εν μέρη ξεκίνησε η τεχνική συζήτηση αλλά θα συνεχιστεί γιατί είναι ένα θέμα που δεν είναι και ασήμαντο αφορά μεγάλο κομμάτι του κλάδου. Δύο ισπανικές τροπολογίες προτείνουν καινούργια κατηγορία και σήμερα το πρωί είπαμε ότι δεν θέλουμε αυτή την καινούργια κατηγορία. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του καταναλωτή όσον αφορά το τι είδους κρασί είναι, αν υπάρχει αναλογία κατηγορία. Και η ενημέρωση μπορεί να γίνει με αναφορά της ανάλυσης του περιεχομένου. Πάντως είπαμε ακόμα αυτό και δεν έκλεισε. Συζητήθηκε σήμερα το πρωί δεν το για να το προσέξουμε περισσότερο. Κάτι άλλο επίσης πολιτικά φορτισμένα. Άρθρο 81. Έχουμε συζητήσει, αλλά δεν έχουμε κρίνει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι θα γίνει με το Λαμπρούσκο ως ποικιλία. Και αυτό θέλει συζήτηση γιατί αφορά πολύ κόσμο. Επίσης και το 93 για την ονομασία πρόλευσης. Θα συζητηθεί κι άλλο να δούμε τι θα γίνει με κάποιες ποικιλίε ε, του, του, του, του σταφυλιού αυτού του Λαμπρούσκο και να δούμε αν θα καλυφθούν όλα τα κρασιά και τα κρασιά που έχουν ή δεν έχουν ενόπνευμα. Σε κάποια σημεία συμφωνούμε. Τώρα για την ετικετοθεσία συζητήθηκε από πλευρά Επιτροπής Περιβάλλοντος για να υπάρχει σύμφωνα με το 119 κάποια υποχρεωτική μνήμα στην ετικέτα. Άρα εκεί δεν έχουμε διαφωνία με την ένβη. Το ψηφίσαμε σήμερα. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι τώρα. Οπότε να υπάρχει αναφορά των περιεχομένων σύμφωνα με αυτό το άρθρο. Τα συζητήσαμε σήμερα. Θα συνεχιστεί η συζήτηση για να δούμε τι θα γίνει με την αναφορά αυτών των ε, στοιχείων του περιεχομένου τώρα για τη θέσπιση νέας κατηγορίας κρασιού για κάποιο κρασί που εν μέρει εν όλο να μην έχει νόμνευμα είπαμε θα το συζητήσουμε κι άλλα τώρα όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών είναι το άρθρο 152, συζητείται στην τεχνική ομάδα. Τώρα για την ποιότητα δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Συζητήθηκε στην τεχνική ομάδα. Και υπάρχει η ένδειξη γραφικής προέλευσης προστασία της ονομασίας, προβλέπεται η καταχώρηση ένα μητρό και οπότε έχουμε κάποιες ε, ε τροπολογίες που δεν θίγουν όμως την ουσία. Σε αυτή τη φάση βρίσκονται επομένω οι εργασίες μας όσον αφορά την κοινή οργάνωση αγοράς. Ευχαριστούμε κύριος Νταντά. Για τρία λεπτά παρακαλώ. Τα περίπου όλα ο εισηγητής, οπότε θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι ένα κείμενο που διορθώνει μετά το Omnibus. Πρόκειται για τα πιο ακαθόδη ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κρασί. Είναι αλήθεια το λαμπρασκά. Και κάθε πολιτική ομάδα συζητάει με τον κλάδο για να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Και η διακοινοβουλευτική ομάδα για το κρασί μπορεί να βοηθήσει επίσης. Κατά τα άλλα δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά που είπε ο συγητής. Πρόεδρος. Ωραίο. Αποκλείεται τόσο γρήγορα η κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα θέλω να ρωτήσω. Εμείς, όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, πάντα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δουλεύουμε βέβαια επικοδομητικά. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και χρησιμοποιούμε σαν βάση τον κανονισμό Omnibus. Τώρα μιλάμε για άλλα προγράμματα στρατηγικής για τα σχολεία κτλ. Μπορούμε να επανέλθουμε γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις στις πολιτικές ομάδες. Και μπορούμε λοιπόν να αξιολογήσουμε ανάλογα με το βάρος που δίνει και το κάθε κράτος μέλος. Επίσης, συμφωνούμε σε ό,τι αφορά τα κρασιά α, χωρίς ή με μειωμένο ενόπνευμα, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει σχετική αγορά και ότι θα πρέπει τελικά ο καταναλωτής να αποφασίσει κατά πόσον θέλει να αποφασίσει να αγοράσει ένα τέτοιο προϊόν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αλλεργίες, για παράδειγμα, και σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να καταναλώσουν αλκοόλ. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι μπορούμε να αποδεχτούμε προϊόντα με μειωμένη υπηρεκτικότητα σε αλκοόλ ή χωρίς ε, αλκοόλ. Για τα άλλα θέματα σε ό,τι αφορά τι απαγορεύσει κτλ. Θεωρούμε ότι έχουν νόημα όλα αυτά, γιατί πρόκειται ίσως και για κάποιες ε, παλιές ε, ε, περιπτώσεις ό,τι αφορά τέτοιες εκτροφές. Γι' αυτό λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, να ευχαριστήσω και για την καλή και επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βιέγας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Γενικώ, πιστεύουμε ότι η στρατηγική κατεύθυνση είναι εσφαλμένη σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση αυτή και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι η λογική να αντικατοστεθούν τα κρατικά συστήματα με μια αυτορύθμιση δεν θα λειτουργήσει στη γεωργία. Να υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο κολεκτιβιστικό μοντέλο και να σπρώξουμε τους ε, αγρότες μας προς την κατεύθυνση αυτή και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, ε, θεωρώ ότι δεν θα είναι βιώσιμο. Τελικά θα οδηγήσει μόνο σε πλεονάσματα και αστάθεια σε ό,τι αφορά τη, τις χώρες. Σε ό,τι αφορά το γάλα και τον τερματισμό των ποσοστώσεων. Είδαμε τι έγινε. Εκατοντάδες ευρώ ε, χρειάστηκαν για να σταματήσουν ε, την πτώση των τιμών. Και στην τελική ανάλυση επικεντρωθήκαμε στις ε, χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης και παραμελήθηκαν οι χώρε τη ε, νότια Ευρώπη, για παράδειγμα στι Αζόρε. Ήταν πολύ σημαντικό προϊόν παραγωγή το γάλα. Είμαστε λοιπόν επί τη αρχή κατά τη ε, περαιτέρω απελευθέρωση της ε, πολιτικής ό,τι αφορά για παράδειγμα την ιδιοπία και την καλλιέργεια. και η απελευθέρωση, για παράδειγμα, για την παραγωγή διαφόρων ειδών ε, κρασιού. Θέλουμε λοιπόν να αντιτηρηθούν οι παραδοσιακές καλλιεργίες για να αντιτηρηθεί η ευρωπαϊκή υπεραξία. Για παράδειγμα, το είδος λαμπρούσκα που επίσης παράγεται στις Αζόρες στο νησί Πίκο, θα πρέπει να συνεχίσετε να παράγεται στις ε, περιοχές όπου υπάρχει παράδοση. Ωστόσο, θα θέλαμε να βοηθήσουμε στην ενίσχυση των εργαλείων που μπορούν τελικά να αποβούν προς όφελος των καλλιεργητών σε μια κατάσταση ενισχυμένης ε, ανταγωνιστικότητας που θα προκύψει αν ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αγορά τη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν αντίστοιχα εργαλεία προκειμένου να αποτραπεί η πτώχευση των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος, νομίζω ότι ο καλύτερο τρόπο για να υποστηρίξουμε τον τομέα τη συνοπία είναι να καταναλώνουμε είναι Η κυρία Χράνς Γκαρσία. Eh, Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο όσο περισσότερο τόσο καλύτερο και όσο καλύτερη ποιότητα ακόμα καλύτερα. Λοιπόν θέλω να πω στον κύριο Αντρέου ότι με απασχολεί ακριβώ το θέμα του ίνου. Και είναι πολύ σημαντικό οι άδειε για καλλιέργειες. Ξέρετε ότι προσπάθησα για παράταση μέχρι το 2050, δεν ξέρω αν έχουμε προχωρήσει καθόλου. Με απασχολεί επίσης το, τα κρασιά χωρίς αλκοόλ. Είναι μια ευκαιρία για εμπόριο στον κλάδο. Να είναι ανοιχτή αυτή η δυνατότητα. Ο ίνος ποιότητας με τις γεωγραφικές ενδείξεις, ε, προέλευση κτλ. Ε, επιβεβαιώνονται έτσι, αλλά η αγορά ζητάει τέτοιου είδου προϊόντα και αν δεν το κάνει αυτό ο κλάδος ο εινοαμπέλικος, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν άλλες εταιρείες που κανονικά δεν παράγουν κρασί αλλά άλλα ποτά και θα ασχοληθούν με αυτό το κλάδο. Είναι σαν να κλέβουν κατά κάποιο τρόπο τη δυνατότητα του αμπελονικού τομέα να μπορέσει να προσθέσει και αυτό το προϊόν στο εμπόριό του. Αυτά είναι που με απασχολούν. Ε, το κρασί χωρίς συνόπνευμα και οι άδειε που δίνονται για δικαίωμα φύτευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Αναφέρεται ότι υπάρχει νέο πεδίο εφαρμογή για τη CMO και για την ΚΟΑ. Και χαίρομαι που περιλαμβάνεται και το χείριο και το κρέας πληρικών Και που τηρείται για τα δικαιώματα καλλιέργειας. Να τονίσω τρία σημαντικά ερωτήματα στο, σημείο αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί ξέρονται τα ιατρικά βότανα από την ΚΟΑ. Είναι σημαντικά αυτά τα προϊόντα. και θα πρέπει να καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογιστικό. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την προστασία των ε, ποικιλιών κρασιού, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει οποιαδήποτε αξιολόγηση για την αγορά, ή για το πώς αυτό θα επηρεάσει τα προστατευόμενα, τις προστατευόμενες ε, καλλιέργειες και τα προστατευόμενα προστατευόμενα είδη κρασιού. Να σας ενημερώσω ότι χθε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας απέριψε την πρόταση αυτή να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αυτό τα κρασιά, τα προστατευόμενα κρασιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον μπορούμε να προστατέψουμε από την χρήση ενός τέτοιου όρου αν ε, ο όρος περιγραφής καλύπτει περιφέρεια και των δύο κρατών. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εξήγηση. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ε, ο κύριος Ντόρφμαν. Ήμουν εισογητής για την γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό και σήμερα το απόγευμα ψηφίσαμε μόλις. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι κάναμε όλη τη δουλειά μας ε, από πλευρά τη Επιτροπή Γεωργία. Πραγματικά εδώ υπάρχουν κάποια σημεία τα ανέφερε και ο εισηγητής ε, που είναι, επιτροπή, που είναι αρμοδίτητα της Επιτροπής Περιβαλλοντικών Υποθέσεων σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ετικετοθεσία για την περιεκτικότητα και τη σύνθεση των κρασιών. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω να αναλάβει την, να αποδεχτεί την θέση μας η Επιτροπή Γεωργίας. Να πω δύο λόγια για την ψηφοφορία. Πιστεύουμε ότι η επισήμανση των θερμίδων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετικέτα Δεν έχουμε προβλέψει όλα τα συστατικά. Και το θέμα των μετουσιωμένων ίνων θα πρέπει να το εξετάσουμε γιατί αποτελεί μια αγορά. Και εγώ, όπως και η κυρία Εράνς Γκαρσία είπε προηγουμένως, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση προέλευσης. Θα πρέπει να υπάρχει νομικό πλαίσιο όμως τα προϊόντα αυτά τελικά. σε ό,τι αφορά τώρα των ε, ινοκαλλιεργητών, δεν μπορούμε. Υπήρξαν κάποιες απαγορεύσεις ε, καλλιεργίας κάποιων προϊόντων για λόγους αλλαγής του κλίματος, ε, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις αυτά τα είδη είναι πιο ανθεκτικά στο κρύο και όχι στη ζέστη. Για τις νέες όμως ε, καλλιεργίες, τα νέα είδη θα πρέπει να είμαστε πιο γενναιοδορείς όπως το λαμπρούσκα. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα είδη τα οποία είναι ανθεκτικά σε διάφορα σε διάφορες συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να επιδείξουμε κάποια παραπάνω υγιεινοδορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις και μία έκκληση. Η παρέμβαση θεωρούμε ότι αποτελεί απαραίτητο μέτρο. Αυτό εκφράστηκε. Αλλά οι μηχανισμοί παρέμβασης θα πρέπει να λειτουργούν πιο γρήγορα. Δεν θέλουμε να κάνουμε ανακοινώσει κτλ. Θα θέλαμε ιδανικά να ισχύουν όλα αυτά από χτε, γιατί ουσιαστικά υπάρχει η χρήση των θέματων αυτών σε ό,τι αφορά την παρέμβαση για τις τιμές κτλ. Κατά δεύτερον, τα προγράμματα για τα λαχανικά και το γάλα για τα σχολεία. Πραγματικά μου προκάλεσε φρίκη αυτά που άκουσα. Σα παρακαλώ λοιπόν να αφήσουμε τα κρατημέλη να εφαρμόζουν όλα αυτά τα προγράμματα χωρί να επιβάλλουμε γραφειοκρατία. Ευχαριστώ πολύ, κύριος... Σαν... κυρία Σάντο. Κύριο Σάντο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο Ρίκ ε, Αντρίου έκανε πολύ καλή δουλειά. Τον ευχαριστώ. Να τον ευχαριστήσω και για τη σημερινή παρουσίαση. Η συνολική εικόνα που μας παρουσίασε θεωρώ ότι είναι σωστή. Είναι σημαντικό να εγγυηθούμε καλή λειτουργία της ΚΟΑ αν θέλουμε να πετύχουμε τους φιλοδοξούς στόχους που θέσαμε για το κλίμα και το περιβάλλον. Αλλά αν θέλουμε επίσης να δώσουμε και μια ευκαιρία να τα βγάζουν πέρα οι γεωργοί. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να πούμε ότι το σχέδιο κανονισμού το οποίο επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνει πολύ μεγάλες μειώσεις το οποίο πραγματικά δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Μιλάμε για μεγάλες ε, ελλείψεις και θα πρέπει να το καταγγείλουμε αυτό, γιατί οι περιοχές με αδύναμες οικονομίες και με με προβλήματα θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά του. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα δεν είναι μόνο η υποστήριξη τη γεωργία. Το θέμα είναι να υπάρχει και μια κάποια εδαφική συνοχή σε αυτέ τι περιοχέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλάνναγκαν. Να πω ότι πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα να προωθήσουμε τον τομέα αυτό με κρασί μετουσιωμένο ή χαμηλής περιεκτικότητας σε, σε αλκοόλ, γιατί και εμένα μου αρέσει το κρασί, μου αρέσει και η λευκή μπύρα, αλλά ξέρω ότι προκαλεί καρκίνο όταν υπάρχει υπερκατανάλωση φυσικά και άλλα πολλά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να τα προωθήσουμε αυτά. Σε ό,τι αφορά τα ιατρικά βότανα, πιστεύω ότι υπάρχει, σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να μπορούν να κινηθούν οι καλλιεργητέ στην Ευρώπη, όχι να επικρατούν τελικά οι εγκληματίε και τα καρτέλ που πληρώνουν τελικά, τα πουλάνε όλα αυτά στα παιδιά σε νοθευμένες μορφές, σε υψηλές τιμές, όπως η κάναβη για παράδειγμα. η αγορά για την ε, ιατρική κάναβη στην Ευρώπη είναι 35,7 δισεκατομμύρια και 49,8 εκατομμύρια η ευρύτερη αγορά. Καλύτερα λοιπόν αυτά τα χρήματα να τα στις τσέπες ε, των γεωργών και να κυκλοφορούν στις κοινωνίες, στις κοινότητές μας και όχι να είναι στα, στις των εγκληματιών που τα ξοδεύουν σε γιότ και πολυτέλειες. Ε, ίσως λοιπόν αυτή την οδό θα έπρεπε να ακολουθήσουμε γιατί πραγματικά θα ήταν καταστροφή για τους εγκληματίες ένα τέτοιο βήμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπράβο στον συνάδελφο Έρικ, τον συγητή. Έτσι θα έχουμε μια αυθεντική μεταβολή και μεταρρύθμιση με, ε, τον, για τον κανονισμό τέλο πάντων που αφορά την κοινή οργάνωση της αγοράς. Προχωράμε, θα φτάσουμε στις συμβαστικές διατάξεις, να δούμε τι θα γίνει, πώς θα κινητοποιήσουμε κάποια μέσα, ούτω ώστε να έχει σωστό προσανατολισμό η αγορά και να κινητοποιήσουμε επίσης και το αποθεματικό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές. Δεν υπάρχει ισορροπία. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες, όπως λέει η Επιτροπή, και επίσης παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιο είδους ε, ε, εγγύησεις αυτές πώς θα υποκαταστήσουν όμως την κρατική υποστήριξη και παρέμβαση υπάρχει μέθοδος ή τεχνολογία blockchain για την λειτουργία της αγοράς το ώστε να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Έχουμε και το θέμα της ε, ελέγχου της προσφοράς για τυριά, για το προσούτο και το κρασί. Όσον αφορά ειδικότερα το κρασί, νομίζω ότι το σύστημα της αδειοδότησης για τη φύτευση θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά το 2030. Δεν θέλω αυτό που θέλει η Επιτροπή όσον αφορά την ονομασία προέλευσης. Θεωρώ ότι το κρασί χωρίς αλκοόλ μπορεί να αποτελεί κάτι θετικό. Χωρίς να θίγει το σύστημα της γεωγραφικής προέλευσης. Να αναφέρονται βέβαια και κάποια στοιχεία ε, όπως οι θερμίδες και τα λοιπά ε, συστατικά του γρασιού. Ευχαριστούμε. Σας ακούμε. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον εισήγητη για το έργο του. Έχω λίγα σχόλια για την δημόσια παρέμβαση. Η πρόταση της Επιτροπής καλύπτει μόνο περιπτώσεις. Θα ήταν καλό όμως και με καλύπτει μόνο το μοσχαρίσιο κρέας για παράδειγμα ενώ θα έπρεπε να καλύπτει και το χείριο γιατί ή τα πουλερικά, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που χρειάζονται το ίδιο. Επίσης, για το κρασί χωρίς αλκοόλ πρέπει να ρυθμιστεί αυτή η αγορά. Υπάρχει, πρέπει να ρυθμιστεί γιατί οι καταναλωτές το ζητούν. Τέλος, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ετικέτα έχει αρκετές πληροφορίες ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να διαλέξει αν θα αγοράσει δηλαδή το προϊόν ή όχι η ετικέτα δεν θα πρέπει να επιτρέπει διπλές, διπλά μέτρα και σταθμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ε, το έχουμε ήδη αναγνωρίσει. Ένα λεπτό, κυρία Ζάνοβα. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Όχι, κυρία Σέντρα. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση έχω στον κύριο Άντρια για τις άδειες φύτευσης σε περίπτωση που έχουμε περισσότερα εκτάρια. Εμείς έχουμε βάλει μια τροπολογία ακριβώ σε περίπτωση περιορισμένων εκταρίων να ευνοείται ο αγρότης σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Η εμπορία του αμπελιού στις Αζόρες επιτρέπεται. Στις Αζόρες έχουμε μια ειδική περίπτωση. Ένα αμπέλι που οι κάτοικοι εκτιμούν πάρα πολύ. Και είναι πολύ καλύτερα προσαρμοσμένο αυτό το αμπέλι στις κλιματολογικές συνθήκες που έχουμε στις Αζόρες και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε υπερβολικά φυτοφάρμακα και τέτοια. Για το ποσέι τώρα. Ο Επίτροπος Φερχόγγιν της Αζόρες είχε πει ότι θα αλλάξει η κατάσταση εδώ. Έχουμε έναν κανονισμό που έχει την εξαίρεση. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε με τη σύγκληση της ΠΑΚ τη μείωση. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό εγώ προτείνω αύξηση στο ΠΟΣΕΙ. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία και τους βοηθούς για τη δουλειά τους αυτή τη βδομάδα που ήταν πολύ φορτωμένη. Θέλω να μιλήσω για τα κρασιά χωρίς αλκοόλ ή αυτά από τα οποία έχει αφαιρεθεί το αλκοόλ. Είναι σημαντικό να μην ξεχνούμε τους ε, παραγωγούς μας. Δεν είναι δυνατόν να εμποδίζουμε την παραγωγή τέτοιου κρασιού. Η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί για τα υπόλοιπα κρασιά πάντως με τον τομέα για να καταλάβουμε κατά πόσο τα κρασιά χωρίς αλκοόλ θα μπορούσαν να καλύψουν το πλώνασμα που έχουμε σε σταφύλια. Έπειτα, πώς θα τα ονομάσουμε αυτά. Κάπως διαφορετικά, όχι κρασί. Οπότε για τις ετικέτες δεν θέλω να αναφέρονται τα συστατικά, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει ενημέρωση των καταναλωτών για τις θερμίδες και όχι στην ετικέτα, αλλά σε εναλλακτικέ πλατφόρμες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή και τους σκιώδη συσυγητές που έχουν βοηθήσει. Επί της ουσίας, θα αρχίσω με κάτι που δεν θα σας εκπλήξει, την παρέμβαση, τα μέτρα στήριξης. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο προσανατολισμός της αγοράς και η παρέμβαση θα πρέπει να παραμείνει ως έχει ως δίκτυο προστασίας όπως είναι και τώρα. Εδώ δεν βλέπουμε δηλαδή από τη δικιά μας την πλευρά κανέναν ελιγμό. Αλλιώς ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας. Και μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα, ό,τι και αν αποφασίσουμε δηλαδή στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τα χρήματα θα είναι περιορισμένα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι κάθε δεκάρα που πηγαίνει για την παρέμβαση στην αγορά δεν θα είναι διαθέσιμο για τις άμεσες ενισχύσεις ή για τη στήριξη της υπαίθρου. Όσον αφορά τώρα τους κανόνες για τις οργανώσεις των παραγωγών και τον ανταγωνισμό γενικότερα. Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει με τον κανονισμό Omnibus που τώρα λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο. Και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε αλλαγή. Οπότε ας μείνουμε στα αποτελέσματα του Omnibus, ας αφήσουμε να δοκιμαστεί κάποια χρόνια και μετά να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Για την πρότασή σας τώρα, το πρόγραμμα για τα σχολεία να πάνε στον κανονισμό του στρατηγικού σχεδιασμού, είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση και συζήτηση δικιά μας η εκτίμηση στο εσωτερικό μας ήταν επειδή διαχειρίζεται η Επιτροπή τα προγράμματα αυτά, θα ήταν δύσκολο. Οπότε περιμένουμε να δούμε διατυπωμένη την πρότασή σας, πώς προτείνετε δηλαδή να λειτουργήσει στην πράξη και θα δούμε. Για τα μέτρα διαχείρισης της αγοράς, η διαχείριση γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξορισμού. Οπότε δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μεταφορά τους από τον κανονισμό στο στρατηγικό σχεδιασμό. Για τον Ίνο. Το νέο καθεστώς αδειών που άρχισε να ισχύει το 2014 και εγκρίθηκε το 2013 λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια και έχουμε άλλα 12 προκειμένου να εκπνεύσει. Σύμφωνα με τους σημερινούς κανόνες, καλό θα ήταν να περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει και να αποφασίσουμε αργότερα, λίγο πριν εκπνεύσει και όχι τώρα. για κάτι το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή μετά από 12 χρόνια. Με το κρασί κάθε φορά έχουμε πολύ έντονη και ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα κρασιά χωρίς αλκοόλ. Η πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ε, να υπάρχει περισσότερη ευελιξία, να ψάξει λίγο τις δυνατότητες που υπάρχουν στην αγορά, ώστε να φυτευθούν αμπέλια, τα οποία να είναι πιο ανθεκτικά ή καλύτερα προσαρμοσμένα στις καταστάσεις. Αλλά από αυτού θα έρθουμε αργότερα. Για τις γεωγραφικές ενδείξεις είμαστε υπέρ της πρότασής σας. Οτιδήποτε μας επιτρέπει να απλοποιήσουμε τα περί των γεωγραφικών ενδείξεων για μας είναι θετικό. Η πρότασή σας πάει προς αυτή την κατεύθυνση, οπότε συμφωνούμε και περιμένουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις σας. Και τέλος, για την τελευταία πρόταση του κύριου Φλάνεγκαν δεν μπορώ να αποφανθώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μιλώ κύριο Αντρέα. δεν καταλαβαίνεις και εσύ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλιά τους. Εντάξει, δεν θα κάνω το... θα αναλάβω εγώ το ρόλο των σκιωδών. Και η κυρία Χέρζανς ε, Γκαρθία, θέλω να την καθισχάσω. Μιλάει εκτός μικροφώνου ο κύριος Αντρίου, δεν τον ακούμε καλά. προτείναμε μέχρι το 2050 με αναθεώρηση το 2023 και μία αξιολόγηση κάθε 10 χρόνια. Αυτή είναι η συνενετική πρόταση μεταξύ των σκιωδών. 2050 είπα έτσι με πρώτη εκτίμηση το 2023 και μετά κάθε 10 χρόνια. Αυτός είναι ο συμβασμός στον οποίο καταλήξαμε. Τώρα, επανέρχομαι σε αυτά που θίξατε. Στον κύριο Ερντός. Και στους άλλους για τα προστατευμένα προϊόντα. Δεν καταλήξαμε. Άνοιξε η συζήτηση, αλλά δεν καταλήξαμε. Γιατί υπάρχουν αντιφατικά. Ο κύριος Στόκμαλ τι λέει, ότι δεν υπήρχε έγκριση για τις ποικιλίε ε, Μπρούσκα και Κλίντον. Η απόφαση δεν ελήφθη πάντως. Για την ερώτηση του κύριου Ερντός για τα βότανα. Λαμβάνεται υπόψη στα παραρτήματα που λέει άλλα προϊόντα. Είναι μια ευρία έννοια τα βότανα. Δεν πρόκειται για ένα προϊόν. Δεν έχουμε καταλήξει οριστικά, ο προσανατολισμός μας πάντως είναι αυτός. Δεν τα ξεχνάμε, αλλά είναι στην κατηγορία άλλα προϊόντα. Για το θέμα της μεταφοράς του προγράμματος ε, οποροκυπευτικά. Ακούω τι λέει η Επιτροπή. Αλλά είναι μια περισσότερο πολιτική απόφαση των σκιωδών που ομόφωνα συμφωνήσαμε. Είναι σαν να δίνουμε ένα δώρο στις χώρες μέλη για να αποφασίζουν για το πρόγραμμα οποροκυπευτικά και γάλα στα σχολεία. Εμείς ε, δεν συμφωνούμε. Για τον κύριο Μπούντα, για το κύριο κρέας, υπάρχει ε, το βόλιο, το χείριο κρέας, η συζήτηση δεν έγινε, αλλά είναι στις συμβαστικές τροπολογίες. Και για την κυρία Ριμπέιρο. Καταλαβαίνω τι λέτε. Και σας ευχαριστώ, γιατί έτσι διευκρινίστε περισσότερο η συζήτηση που είχαμε στους κοιόδους εισηγητές. Παρόλο που δεν έχουμε καταλήξει και έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Δεν απελπίζομαι με το ρυθμό και την ε, συλλογική βούληση. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε συμβαστικές τροπολογίες για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν Πρόεδρε και εντάξει νομίζω είμαι στην ώρα μου έτσι μέχρι τις 6.30 δεν είχα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρο, Κυρίες και κύριοι. Υπάρχει διχογνωμία, υπάρχει ποικιλία απόψεων, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, αυτό είναι δημιουργικό και νομίζω ότι ε, όσο συζητήσαμε και στα όσα είπε ο κύριος Αντριέ, ε, καταλήξαμε στο ότι έγινε βήματα προόδου και στο ότι φαίνεται φως στην άκρη τούνελ. Νομίζω ότι τα καταφέρουμε σιγά σιγά και πάλι σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε καλή δουλειά θα τα ξαναπούμε στις 7, κατόπιν στις 18 και 19 Φεβρουαρίου. Και στις 27. Επομένως βλέπουμε ότι ο Φεβρουάριος είναι ο κρίσιμο μήνας για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα στις συνεδριάσεις, οι συντονιστές θα συναντηθούμε στο 4Q2. Δύο ρόγους πιο κάτω συντονιστές στο 4Q2. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς. Πολύ καλή συνεδρίαση.